Good afternoon everybody. Καλώς ορίσατε όλοι. Ελπίζω να χαρήκατε το μεσημεριανό σας διάλειμμα, τουλάχιστον εγώ το χάρηκα και ελπίζω κι εσείς. Τώρα ξέρω ότι είναι δυόμιση ώρα, είναι δύσκολη ώρα για τους ε, συναδέλφους. Θα καταφτάσουν αργότερα οι περισσότεροι. Ε, θα έχουμε και άλλους. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους ε, εξαίρετους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους και όλους συμμετέχοντες. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω ε, για τη στη δημόσια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή ΑΦΚΟ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Αναφοράς, η κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ είναι πρόεδρος της Συνταγματικής και θα έρθει λίγο αργότερα. Καταρχάς θα ήθελα να σας δώσω μερικές πρακτικές πληροφορίες. Έχουμε διερμηνία σήμερα σε όλες τις επίσημες γλώσσες μας, με εξαίρεση τα κροατικά, τσεχικά, εστονικά, ε, λετονικά, λιθουανικά, φιλανδικά και σλοβενικά. Επίσης, ε, ε, παρακαλώ, σημειώστε ότι μεταδίδονται στο διαδίκτυο τα λεγόμενά σας, δηλαδή όταν παίρνετε το λόγο θα απευθύνεστε στους Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα η ακρόασή μας θα ασχοληθεί με την πρόσφατη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για να δούμε σε κατά πόσο ανταποκρίνεται η πρόταση αυτή στις προσδοκίες των ενεχομένων και των Ευρωπαίων πολιτών φυσικά. Όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά, θεώρηση ε, του νομικού πλαισίου έπρεπε να έχει έρθει εδώ και καιρό. Ο κανονισμός που υπάρχει σήμερα γνωρίζει δυσκολίες. Από την πρώτη ε, θέση σε ισχύ του από το 2012 και μετά ε, πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών να βάγισαν ε, στο στάδιο της καταχώρησης. Ακολούθησαν ε, σημαντικές αποφάσεις από ευρωπαϊκά δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται και ερμηνεύεται ε, από πλευρά τη ε, ο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ήταν υπερβολικά αυστηρό και υπερβολικά περιοριστικό καμιά φορά. Οπότε η Επιτροπή μα Αναφορών μαζί με τη Συνταγματική Επιτροπή καλωσορίζουν τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει ε, εκβάθρων ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το νομικό πλαίσιο και το διαδικαστικό για να είναι πιο προσβάσιμη και πιο αποτελεσματική ελπίζουμε για τη συμμετοχή του κοινού ε, στην λήψη των αποφάσεων και χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν ήταν οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις πριν μπούμε στην ουσία και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχηθώ μια συζήτηση πολύ ε, γόνιμη και αποδοτική και ευχάριστη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές. Έχουμε τον κύριο Μάρτεν Χρότ, που είναι συντονιστής της Εκστρατείας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Έχουμε την κυρία Λίσα Λιρόνη από το Κέντρο Υποστήριξης και τον κύριο James Όργαν που είναι λέκτορας δικαίου στη νομική σχολή ε, του Λίβερπουλ. Νομική σχολή και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεχρότ ε, από τη ΜΚΟ ε, Εκστρατεία Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Θα σας παρακαλούσα όλοι να τηρήσετε αυστηρά το χρόνο σας, 10 λεπτά έκαστος. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Ντεχρότ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε. Μάρτιν Ντεχρότ και είμαι στις Βρυξέλλες από το ECI Campaign. 15 ετών είναι η ΜΚΟ μας με αποκλειστικό στόχο να πετύχει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για πρώτη φορά στον κόσμο βλέπουμε μια δημοκρατία συμμετοχική, ηλεκτρονική, ηλεκτρονική διευκόλυνση δηλαδή. Ε, χαιρόμαστε που οι ευρωβουλευτές πίεσαν καταρχάς να εγγραφεί στη συνθήκη αυτό το μέσο και στη συνέχεια να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι όλα ρόδινα για να μην πω τίποτα χειρότερο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Θέλουμε και ε, για άλλη μια φορά να στραφούμε όπως και στο παρελθόν προς εσάς στο Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσετε γιατί ψυχοραγεί ε, με αργό και οδυνηρό θάνατο απειλείται η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αυτό είναι μια άμεση εντολή από τους Ευρωπαίους πολίτες και κρίσιμο. Είναι εξαιρετική ευκαιρία η πρωτοβουλία πολιτών για να κάνετε εσείς μια ε, συζήτηση και να συνεργάζεστε με τους Ευρωπαίους ε, πολίτες ε, ανάμεσα σε δύο ευρωεκλογές. Και η ίδια η πρωτοβουλία σας χρειάζεται να την κάνετε περισσότερο κτήμα σας για να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει και στο μέλλον. Στην παρουσίασή μου καταρχάς θα σας παρουσιάσω ε, τι ε, πιστεύουμε ότι διακυβεύεται. Μετά θα σας πω πώς αξιολογούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέλος θα σας κάνω και προτάσεις για τη διαδικασία αναθεώρησης και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχίζω από το πρώτο. Τι διακυβεύεται τώρα κατά την περίοδο αυτή, κατά την άποψή μας, περίοδο αναθεώρησης. Σας δώσω κάποια στοιχεία έτσι χοντρικά. 69 πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταχωρίστηκαν 48 και μόνο 4 πρωτοβουλίες έχουν ξεπεράσει το κατόφλι του 1 εκατομμυρίου υπογραφών για να γίνουν παραδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μιλώ μόνο για τις υπογραφές. 8 με 9 εκατομμύρια υπογραφές έχουμε συλλέξει. Τα 2 τρίτα, ίσως και παραπάνω, ε, των υπογραφών αφορούν τις τέσσερις επιτυχείς εντό εισαγωγικών ε, πρωτοβουλίες που ευωδόθηκαν. Και οι μισές ε, κατά τη διάρκεια της έναρξης εφαρμογής το 2013 και τα τελευταία τέσσερα χρόνια μία ήταν η σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας βλέπουμε λοιπόν ε, αυτές τις τέσσερις πρωτοβουλίες να κυριαρχούν. Δύο πρωτοβουλίες απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καμία δικαιολογία. Οι δύο πρωτοβουλίες, One of Us και άλλοι, να σταματήσουν τα πειράματα στα ζώα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες προτάσεις σε σχέση με το δικά μας το νερό Ωστόσο, αυτά είναι αυτά που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση από τους ε, διοργανωτές το δικαίωμα στο νερό ήταν η μία και το άλλο σταματήστε τη γλυφοσάτη. Ε, δεν είναι τα ίδια διοργάνωτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και στι πολύ λίγε περιπτώσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ανταποκρίθηκε θετικά, οι διοργανωτέ είναι δυσαρεστημένοι. Σα δείχνω εδώ τι λένε ότι προσπαθεί να μας σταματήσει την πρωτοβουλία ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες ασαφείς και θολές προτάσεις ε, περί διαφάνειας. Από τη μια ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι επιτυχία και ότι ακούει τους πολίτες και από την άλλη οι διοργανωτές και εκείνοι που μαζεύουν τις ε, υπογραφές έχουν τελείως διαφορετική εικόνα και αντίληψη για την επιτυχία αυτή. Έρχομαι τώρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε εδώ αυτή τη διαφάνεια όπου αναγράφονται οι 12 ε, μεταρρυθμίσεις ή καλύτερα τα αιτήματά μας για μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία είναι πάγιο αίτημά μας ε, και έχω βάλει και διάφορα χρώματα ανάλογα με το ποια αιτήματα έχουν αντιμετωπιστείτε από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε από τη δράση της μέχρι τώρα. Όπως βλέπετε έχουν καταβληθεί ε, σημαντικά βήματα και προσπάθειες για να γίνει πιο φιλική προς το χρήστη αυτή η πρωτοβουλία. Αν δείτε όμως το σημείο 2 και 3, ε, τον πολιτικό αντίκτυπο, τα πιο βασικά πολιτικά ζητήματα δεν έχουν λυθεί. Πόσο μάλλον αντιμετωπιστεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον υπόλοιπο χρόνο μου θα ήθελα να επικεντρωθώ λοιπόν σε αυτά ε, τα σοβαρά που λείπουν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την άποψή μας. Το πρώτο θέμα το πεδίο που ε, καλύπτει η Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει στο Συμβούλιο ε, αναθεώρηση των συνθήκων και η Πρωτοβουλία των Πολιτών αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θυμάστε την απόφαση του δικαστηρίου σταματήστε το TTIP ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ερμηνεύει αυτά με την ευρία έννοια και να κάνει πρόταση στο Συμβούλιο τροποποίησης αναθεώρησης των συνθήκων. Όπως απεφάθηκε το ότι, ότι, το δικαστήριο, συγγνώμη, ότι πρέπει ένα αντίστοιχο νομοθέτημα να υιοθετηθεί. Και μόνο έτσι θα αναπτυχθεί πλήρως και θα πιάσει τόπο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δηλαδή να γίνεται μια συζήτηση σε όλα τα κρατημέλη για μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Ένα άλλο θέμα και σε σχέση με αυτό που είπα προηγουμένως έχει να κάνει με το εξή. Τι γίνεται με τη συνέχεια και την παρακολούθηση που γίνεται και ποιο ερώτημα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς μπορεί κανείς να δικαιώσει αυτούς τους πολίτες που έχουν κινητοποιηθεί με τόση ενέργεια και τόσο κόπο και πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό στην πράξη ώστε να πιάσει πολιτικά τόπο. Κυρίως ε, στρεφόμαστε προς εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από εσά περιμένουμε να παίξετε ε, ρόλο πρωταγωνιστικό για τη συνέχεια που, που δίνεται στις επιτυχείς ε, πρωτοβουλίες θα πρέπει να παρακολουθείτε με έκθεση κάθε επιτυχή πρωτοβουλία πολιτών, να λέτε τι ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το ψηφίσετε στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που δίδεται στις ε, επιτυχείς και παραδεκτές πρωτοβουλίες. Επίσης, και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως έδειξε η πρωτοβουλία για τη γλυφωσάτη, αυτά όλα έγιναν ερήμην ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι που μας εκπλήσει πάρα πολύ. Ε, τελικά τα κράτη-μέλη μπλόκαραν το σημαντικότερο αίτημα που ήταν η απαγόρευση της γλυφωσάτης. Και η απόφαση αυτή ελήφθη πριν ε, εκδοθεί η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό λοιπόν και κρίσιμο να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, άρα και δια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ας πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να συμμετέχει σε δημόσια ακρόαση και να καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετέχουν και στην αξιολόγηση. Όχι υποχρεωτικό, αλλά να προσκαλούνται. Στη συνέχεια, οι επιτυχίες ε, πρωτοβουλίες πολιτών είναι μειονότητα, δηλαδή εκπροσωπούν μειονότητα Ευρωπαίων πολιτών, παραμένει μειονότητα. Θα πρέπει όμως να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις ε, γνωμοδοτήσεις, τις εκθέσεις θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται για τις δραστηριότητε αυτές, τις πρωτοβουλίες, τις εκθέσεις ε, και να υπάρχει μια δημογραφική ισορροπία στην παρουσία στις Βρυξέλλες ε, για να ενημερώνονται για τα υπέρ και τα κατά τους περιορισμούς μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών που έχει κριθεί παραδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, η πολιτική ε, λογοδοσία θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί στο στάδιο της καταχώρησης Έχουμε ένα μηχανισμό λογοδοσίας, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάνει τη νομική αναθεώρηση, υπάρχει αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε προβλέπεται, στο τέλος της, του κύκλου ζωής της πρωτοβουλίας. Ωραία, εγκρίνεται, ε, θεωρείται παραδεκτή και αν έχουν κάποιο πρόβλημα είναι δυσαρεστημένοι οι ε, διοργανωτές και οι εμπνευστές δεν έχουν που να καταφύγουν στο δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει άλλη μια δημόσια ακρόαση μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει την απόφαση της και να την τεκμηριώνει και οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, Ευρωβουλευτές και άλλοι ενδεχομένως ενεχόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπολείπους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρίβεια των λόγων σας και την ακρίβεια επίσης του χρόνου. Ελπίζω να δώσετε το καλό παράδειγμα και να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να συμμετέχουν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. αργότερα. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ελίσσα Λιρώνη. Παρακαλώ. ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή ε, η Υπηρεσία Δράσης Πολιτών, την ΕΚΑΣ. Λέγομαι Λίσα και είμαι ε, διαχειριστής ψηφιακής δημοκρατίας ε, για την ΕΚΑΣ που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στις Βρυξέλλες και που εδώ και 27 χρόνια δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα από τα δικαιώματα των πολιτών βεβαίως είναι και η συμμετοχή στη ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. Σήμερα θα σας παρουσιάσω λίγο την άποψή μας ε, για τον κανονισμό. Τι θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικό για μας, ε, ποια στοιχεία ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να εγκριθούν και κάτι παραπάνω για την παρακολούθηση και τον αντίκτυπο αυτών των πρωτοβουλίων των πολιτών. Καταρχάς η ΕΚΑΣ όπως και το ECI Campaign, ε, είμαστε από την αρχή που εγκρίθηκε αυτό το εργαλείο, προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το μοναδικό ε, διεθνές εργαλείο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζουμε μαζί με άλλες δύο οργανώσεις, το Democracy International και την, ε, το ε, Ινστιτούτο Πρωτοβουλειών. Ε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ε, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους διοργανωτές των πρωτοβουλειών ε, των πολιτών με τρεις τρόπους. Ε, νομικές συμβουλές πριν υποβάλουν την πρότασή τους, ε, συμβουλές για την εκστρατεία και την επικοινωνία μέσω της Democracy International και τους δίνουμε και τις δυνατότητες να μεταδίδουν ζωντανά στα μέσα επικοινωνίας αυτές τις συμβουλές και να ενισχύουν το δίκτυό τους. Επίσης η ΙΚΑΣ ήταν υπεύθυνη για τις νομικές συμβουλές, δωρεάν υπηρεσίες αυτές για τους πολίτες και ε, χρησιμοποιώ τον αόριστο ε, διότι αυτή τη στιγμή η ΙΚΑΣ είναι σε μια κοινοπραξία που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της νέας διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για φέτος και στο τέλος της παρουσίαση θα σας εξηγήσω λίγο γιατί θεωρούμε ότι είναι ε, μια σημαντική υποστηριστική υποδομή. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω μια σύντομη εικόνα των διαφόρων σημείων που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά στην αναθεώρηση και πρέπει να πούμε ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άσια Κοβρακόβα, η Διευθύντρια, ε, μας το 2016 έστειλε μια γνωμοδότηση ως τμήμα της πλατφόρμας για βελτίωση της πρωτοβουλίας πολιτών. Αυτή η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή τότε στην πλατφόρμα του Refit ως ε, μία από τις επίσημες γνωμοδοτήσεις ε, και ε, συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα του εργασίας του 2017. Όσοι δεν γνωρίζετε την πλατφόρμα Refit, ε, ε, είναι κάτι το οποίο συστάθηκε στη διάρκεια της πρότασης και της ανακοίνωσης για την καλύτερη νομοθεσία και αρμόδιος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Τίμερμανς. Και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έλαβα υπόψη του έξι σημεία τα οποία είχαμε προτείνει για βελτίωση της πρωτοβουλίας πολιτών. Τα μόνα σημεία με τα οποία δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι είναι στο πρώτο θέμα, το θέμα ε, της δοκιμής της ε, νομικής αποδοχής, κατά πόσο είναι παραδεκτό κάτι. Ε, στο τελευταίο σημείο επισημαίνουμε ότι υπάρχει πίεση για περισσότερες νομικές συμβουλές, αλλά αυτό το οποίο δεν μας καθησυχάζει και πάρα πολύ είναι ότι ακόμα δεν είναι απόλυτα σαφές, σαφές ε, τι σημαίνει ε, ότι είναι εκτός της ε, εξουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάποιες νομικές πράξεις και το πώς ορίζονται. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η διατύπωση αυτή μπορεί να βελτιωθεί για να βοηθήσει και τους διοργανωτές να καταλάβουν καλά τι μπορούν να προτείνουν και τι δεν μπορούν να προτείνουν. Τώρα, όσον αφορά τις απαιτήσει των δεδομένων, θεωρούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι Διότι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους οι διοργανωτές ε, των πρωτοβουλειών είναι απογοητευμένοι με αυτό το εργαλείο είναι γιατί ε, δυσκολεύονται να το χρησιμοποιήσουν, οι πολίτες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση και τώρα πιστεύουμε ότι απλουστεύοντας και εναρμονίζοντας τι τις απαιτήσεις δεδομένων και Εγκρίνοντας μια ενοποιημένη προσέγγιση για τη συλλογή των δεδομένων και των εντύπων είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν όλα αυτά. Και επίσης στην πρόταση υπάρχει η, η εναρμόνιση των απαιτήσεων δεδομένων και από 13 διαφορετικά έντυπα τώρα θα έχουμε μόνο δύο και υπάρχει η δυνατότητα να επιτρέπουμε στους πολίτες να υπογράφουν βάσει εθνικότητας ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, επομένως υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις απαιτήσει των δεδομένων. Τώρα όσον αφορά το τρίτο θέμα και εδώ μα ικανοποιεί το γεγονός ότι οι επιτροπέ πολιτών είναι κάτι το οποίο ε, προβλέπεται, δηλαδή οι διοργανωτές θα μπορούν να ε, καθορίσουν ότι αυτές οι επιτροπές πολιτών είναι νομικά πρόσωπα και επομένως ε, αυτό είναι μια βελτίωση για μας. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση με την περίοδο συλλογής υπογραφών των 12 μηνών. Ένα χρόνος δεν αρκεί για να συλλέξουμε ένα εκατομμύριο ε, υπογραφές 28 διαφορετικά κράτη-μέλη. Επομένως, εμείς προτείναμε είτε να παρατηθεί η περίοδος αυτή στους 18 μήνες ή να υπάρχει ένα διάστημα ε, μεταξύ της ε, ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας που μπορούν να αρχίσουν να συλλέγουν υπογραφές και όντω η Επιτροπή δέχτηκε αυτό το τρίμηνο και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το προχωρήσει αυτό. Το πέμπτο είναι η διαδικτυακή συλλογή υπογραφών και όπως θα είδατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 2020 να υπάρχει ένας μόνιμος ελεύθερος σερβερ στη διάθεση των διοργανωτών πρωτοβουλειών των πολιτών και δεν θα υπάρχει ανάγκη για πιστοποίηση του διαδικτυακού συστήματος συλλογής από την ε, στις εθνικές αρχές. Επομένως αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να το προωθήσουμε. Και τελευταίο, ε, εκστρατείες ενημέρωσης ε, της πρωτοβουλίας πολιτών. Εδώ και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο όσον αφορά την ύπαρξη του συγκεκριμένου εργαλείου, αλλά και για να βοηθήσουμε τους διοργανητές ε, να ε, τους δίνονται περισσότερες κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει να εγκριθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Ο συνάδελφος ο Μάρτιν ε, που μας είπε ότι το βασικό ε, πρόβλημα και η απογοήτευση των πολιτών ε, προκύπτει κυρίως λόγω της συνέχειας που δίνεται στην πρωτοβουλία των πολιτών. Η δική μας η συμβουλή ως ΕΚΑΣ είναι ότι ναι μεν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνει αλλαγή της συνθήκης και από τη συνθήκη είναι σαφές ότι οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν, να καλέσουν την Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό το να καλέσουν είναι η ουσιαστική ορολογία. Δεν μπορούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναλάβει πρωτοβουλία για μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Ε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν όρισε ακριβώς ε, τι είναι νομική πράξη, legal act και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυφθούν. Θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο μορφές νομικής πράξης. Η μία είναι νομικά δεσμευτικά ε, μέσα, τα οποία βέβαια πολύ δύσκολα μπορούν να προσεγγίσουν οι πολίτες, ε, ε αν λάβουμε υπόψη ότι ούτε καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πρωτοβουλία για νομοθετικές προτάσεις. Επομένως, για μας είναι πολύ δύσκολο με ένα εκατομμύριο υπογραφές να μπορούν οι πολίτες να ε, αναλάβουν πρωτοβουλία για μια πρόταση. Αλλά υπάρχει άλλη δυνατότητα για τις άλλες νομικές πράξεις που είναι ε, μη νομικά δεσμευτικά μέσα, αλλά είναι συστάσεις και γνωμιδοτήσεις οι οποίες προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πιστεύουμε ότι ίσως ε, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει θέσει υποχρεωτικά μη νομικά δεσμευτικά μέτρα, ε, το οποίο δίνει ένα μήνυμα ότι ίσως αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών θα μπορούσαν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τα θεσμικά όργανα. Και δεύτερον, συμφωνώ με τον Μάρτιν, διότι και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις ε, πρωτοβουλίε των πολιτών που φτάνουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Ε, πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να διοργανώσει ένα σύστημα ψηφοφορία κάθε φορά που υπάρχουν ένα εκατομμύριο υπογραφέ σε μια πρωτοβουλία πολιτών και να αποφασίζουν συνολικά ω εκπρόσωποι των πολιτών. Και αυτό πιστεύω ότι θα δώσει μια πολύ ε, ισχυρή φωνή και ε, θα φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη ε, οι, οι απόψει του από του ηθήνοντε. Ε, πολύ σύντομα για να ολοκληρώσω, πιστεύουμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη υποδομές υποστήριξης για τους διοργανωτές των πρωτοβουλειών και εδώ, όπως σας έλεγα, υποστηρίζουμε την πρόταση για τη διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πριν περάσω στην επόμενη διαφάνεια πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εν γέννη θα πρέπει πάντα να έχουν κατά νου ότι οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών υπάρχουν για να ε, δρουν ω ενδιάμεσο μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και στόχο μα είναι να υποστηρίζουμε τα ευρωπαϊκά ε, ε, θεσμικά όργανα. Ορισμένε φορέ είμαστε επικριτικοί μεν, αλλά προσπαθούμε όντω να δρούμε ω ενδιάμεση, να εξηγήσουμε στου πολίτε ότι κάνετε καλή δουλειά και εμεί απλώ προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να σα πλησιάσουν. Και κάτι τελευταίο, μια τελευταία διαφάνεια για την πλατφόρμα αυτή τη συνεργασία ε, για να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να στηρίξει. Η πλατφόρμα θα είναι μια ε, πλατφόρμα ε, στην οποία οι πολίτες ε, και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας μπορούν να μάθουν περισσότερα για μια πρωτοβουλία. Θα μπορούμε επίσης να συζητήσουμε την πρόταση, να βρούμε δίκτυα στην Ευρώπη στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον και να συνεργαστούμε μαζί τους και να υπάρχουν και πρωτοβουλίες επιτροπές πολιτών και θα υπάρχει επίσης και κάτι το οποίο γίνεται ανεπίσημα, θα υπάρχει ένα γραφείο δίκτυο στήριξη που θα δίνει νομικέ συμβουλέ, συμβουλέ για τι εκστρατείε και επικοινωνία και έτσι θα έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να υποβάλουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ενημερωτικά αυτά που μας είπατε και σήμερα ο τρίτος ομιλητής είναι ο James Organ ο οποίος είναι ε, καθηγητής ε, δικαίου και κοινωνικής δικαιοσύνης στο Λίβερπουλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ε, και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, αλλά υπάρχει το θέμα της συνέχειας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αξίζει συγχαρητηρίων που έχει εισαγάγει αυτό το εργαλείο, ε, το ECR, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Συγχαρητήρια και στο Κοινοβούλιο. Αυτά όσον έχει στο νομικό πλαίσιο, βεβαίως χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, και πέρα από την πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί. Θα προσπαθήσω να δώσω μια νομική χρειά σε κάποια από τα σχόλια τα οποία έκαναν οι δύο προλαλήσαντες. Να ε, σχολιάσω τους ε, στόχους ε, και να πω, να αναφερθώ στις περιπτώσεις επί των οποίων έχουμε λάβει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Ελπίζω όλα αυτά να βοηθήσουν τη συζήτηση. Ας δούμε τι είναι το ECI. Το ECI πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το εξή. Το ECI είναι σημαντικό για να υπάρχει η δημόσια συζήτηση, αλλά υπάρχει και ένας ε, δεύτερος σημαντικός ρόλος, η εφαρμογή της πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το άρθρο 11.4 και ο σχετικός κανονισμός. Και είναι αυτό το δεύτερο ε, το οποίο δίνει στο ECI την ε, δημοκρατική του ισχύ και ξεχωρίζει το ECI από άλλες ε, μορφές συμμετοχής των πολιτών, κυρίως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 11. Το θέμα της επιρροής είναι ιδιαίτερα επίμαχο κυρίως όσον αφορά τις ε, αλλαγές ε, σχετικά με το ECI. Αν δούμε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος, ο στόχος είναι να διερωτηθούμε κατά πόσο οι πολίτες θα ε, χρησιμοποιούν το ECI για να υπάρχουν περισσότερες συζητήσεις ή κατά πόσον θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ECI έτσι ώστε να υπάρχει άμεση και συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ένας από τους στόχους είναι η μεταρρύθμιση ε, να είναι ε, πιο εφικτή, ε, πιο λειτουργική και θα τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Βεβαίως η έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή είναι η νομική, οι νομικές πτυχές του θέματος. Η καταγραφή η καταγραφή θα πρέπει να είναι όσο πιο ευρία γίνεται. Όπως αναφέρεται στην περίπτωση Κωνσταντίνη, εγώ ε, θεωρώ ε, μια περιοριστική ε, ερμηνεία του ECI, αυτό θα περιορίσει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Η διαδικασία καταγραφής πρέπει να είναι απλή τα ECI ε, μπορούν να ε, καταγράφονται ε, το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει το ρόλο του θεσμικού μέντορα για τα ECI ή κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει περισσότερο ένας ανεξάρτητος φορέας. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι το ερώτημα του, της σύγκρουσης που μπορεί να υπάρξει. Ε, όπως βλέπουμε και με το TTPCI υπάρχουν και κάποιοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο να μην θέλει κανείς να καταγράψει την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το θέμα αυτό είναι νομικό ε, και δεν θα πρέπει κανείς ε, να εξετάσει την ουσία των θεμάτων. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα του, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, το πιο εύκολο είναι να έχουμε έναν ανεξάρτητο φορέα ο οποίος θα κρίνει το παραδεκτό και το επιτυπητό της καταγραφής. Όπως ακούσαμε και από τους ε, προηγούμενους ομιλητές, ε, η επόμενη φάση, η φάση υποβολής, είναι και η πιο σημαντική. Η μεταρρύθμιση ε, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και όσον αφορά την εκστρατεία, εδώ υπάρχει μία μεγάλη ευκαιρία ε, να ε, ασχοληθεί κανείς με τις ε, υπογραφές, με την πολιτική. Επίσης είναι και μια ευκαιρία για διαθεσμική συνεργασία σε αυτήν την χάραξη της πολιτικής. Το ECI, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ως εργαλείο πρέπει να υπάρχει η καταγραφή, όπως είπαμε, και εδώ πρέπει να υπάρχει και σχετική συμμετοχή των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας και μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό το δικαίωμα. Ε, καθαρά νομικά είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει νομοθετική πράξη. Το άρθρο 114 λέει ότι η πρωτοβουλία αυτή ε, δεν είναι δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όμως υπάρχουν αρκετές ε, εναλλακτικέ λύσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική επιρροή. Όσον αφορά τον κανονισμό, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρξει κάποια προαιρετική δέσμευση από πλευράς Επιτροπής να ε, θεωρηθεί ότι είναι μία νομική πράξη, μία απάντηση ε, σε ένα επιτυχημένο ECI. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ε, με αυτόν τον τρόπο όμως ε, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το δικαίωμα της ε, πρωτοβουλίας. Αυτές οι προτάσεις οι οποίες σας λέω δεν είναι δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αμφισβητούν το νομικό δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας. Η Κομισιόν μπορεί να προσφέρει την αρνησή της σε μια πρόταση που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Τώρα, το θέμα είναι ότι ε, θα πρέπει ε, οι πολίτες ε, να αναφερθούν λιγάκι στο δικαίωμα της πρωτοβουλίας να μπορούμε βέβαια να έχουμε μια τέτοια παραδοχή. Αυτό σημαίνει ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες και ενισχύει και το ECI. Υπάρχουν εναλλακτικές μορφές συμμετοχής, όπως ακούσατε ήδη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει μεγάλη ευκαιρία να συνδυάσει κανείς ε, τη νομιμότητα δημοκρατικών εργαλείων και ε, την, ε, τον αντιπροσωπευτικό φορέα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί αυτό βοηθάει στην ομοποίηση των συζητήσεων. Κατόπιν υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι δημοκρατικής συμμετοχής, Εάν όλα αυτά προκληθούν από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί κανείς να ελέγξει τις προτάσεις και ο τρίτος τρόπος είναι να συμμετέχουν οι ίδιοι οργανητές ε, στη διαδικασία να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσα από λόμπι για να μπορούν να παραμείνουν και πέρα από ένα επιτυχημένο ECI. Τώρα, όσον αφορά τις ε, προτάσεις ε, για ε, τροποποίηση των συνθήκων. Εγώ νομίζω ότι εδώ αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε ένα νομικό εργαλείο που λέει ναι πράγματι όλα αυτά είναι εφικτά. Βέβαια το εργαλείο δεν είναι απόλυτα σαφές αλλά υπάρχει μια, ένα επιχείρημα ότι η πρωτοβουλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Το άρθρο 48.2 δίνει στην Επιτροπή τη δύναμη ε, τροποποίησης των ε, συνθήκων. Άρα δηλαδή ε, αυτό εμπίπτει τι αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το δεύτερο θέμα είναι κατά πόσον αυτό πρέπει να γίνει με στόχο ε, την ε, εφαρμογή των συνθήκων. Αυτό ε, είναι λιγότερο σαφές, αλλά οι πολίτες μπορούν να πιστεύουν ότι ένα κομμάτι της συνθήκης μπορεί να τροποποιηθεί για να εφαρμόζονται, παραδείγματο χάνει οι αξίε που υπάρχουν στο άρθρο 3. Άρα δηλαδή υπάρχει αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι θα βοηθούσε στο να ενισχυθεί το ECI. Τέλος, θα μιλήσω για κάποια θέματα που έχουν προκύψει στα δικαστήρια. Ευχαριστώ μετά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Έξι περιπτώσεις, οι δύο πιο γνωστές ε, είναι οι περιπτώσεις εκείνες ε, όπου ανετράπει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι περιπτώσεις ε, υπογραμμίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ακούσει σχετικά με τη σημασία, το πόσο σημαντικό είναι να ερμηνεύονται με ευρύτητα οι ε, νομικές περιπτώσεις Έχουμε ακούσει ότι η δημοκρατία είναι εξίσου σημαντική για εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις και δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός. Και επίσης ε, υπάρχει και η δημοκρατική σημασία του ECI κυρίως ε, η υποχρέωση ε, να αναφέρονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Βεβαίως ε, το δικαστήριο είπε ότι η συμμετοχή των πολιτών δεν μπορεί να επηρεάζει την απόδοση εξουσίας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί πάντα να λαμβάνει κάποιες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο αυτής της αρχής. Και θα ήθελα να σταματήσω εδώ, προσβλέπω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ παρόλο που όλοι σα ήσασταν σαφέστατοι, είμαι σίγουρη ότι θα έχουν πολλέ ερωτήσει, οι συνάδελφοι. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Βαλένσα, α πούμε, για αρχή, που είναι ο εισηγητή τη Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. I wonder... Uh, I wonder if... Ε, πρόεδρε, εγώ αναρωτιέμαι αν η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά φιλόδοξη, έτσι ώστε να είναι αρκετά ευέλικτη η διαδικασία αξιολόγησης και ε, έγκρισης ε, για να χαρακτηρίζονται περισσότερες πρωτοβολίες ως παραδεκτές, να καταχωρίζονται ε, και να δίνεται συνέχεια. Αρκεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σκοπό. Έχω και δεύτερη ερώτηση όμως. Υπάρχει μια αντίληψη στον πληθυσμό για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά τη διαδικασία έγκρισης ε, χαρακτηρισμού ως παραδεκτής μιας πρωτοβουλίας και κατά τη συνέχεια δίνεται πολιτική και νομική. Τι λέει ο κόσμος. Ε, θα ήθελα τη δική σας άποψη. Έχω μια ιδέα. Ευχαριστώ από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η συγγετής είναι ο κύριος Σόπφλιν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Sharon. Thank you Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να κάθομαι εδώ στα ψηλά ε, σε αυτές τις ψηλές θέσεις. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. Δεν θα κάνω εγώ όλες τις ερωτήσεις που σκέφτομαι να κάνει και κανένας άλλος. Το πρώτο, αυτό που είπες, James Organ, το τελευταίο, είπε για την πολιτική, για την εφαρμογή πολιτικής, ότι η πρωτοβουλία των πολιτών έχει στόχο αυτό, έχει στόχο να θέσει την ατζέντα. Όχι μόνο αυτό, έχει και την ε, συνειδητοποίηση του κόσμου. Αυτό δεν είναι ρητό, αλλά υπονοείται. Ε, είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού, κουλτούρας, αλλά δεν θα πρέπει να το παραμελούμε. Αν ένας μεμονωμένος πολίτης απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ρωτάει γιατί δεν το έκανε αυτό, είναι άλλο πράγμα και άλλο ειδικό βάρο έχει και βαρύτητα αν μαζέψει και ένα εκατομμύριο ε, υπογραφές. Ε, μετά και στις τρεις παρουσιάσεις σας κατά κάποιο τρόπο αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα ε, του ανεξαρτήτου φορέα που θα πρέπει να ελέγχει το παραδεκτό και να το επαληθεύει. Είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να είναι επιθυμητό από τη σκοπιά της δημοκρατίας θεωρητικά Βεβαίως δεν μπορεί να είσαι κριτής και κρινόμενος. Αυτά είναι βασικά στοιχειώδη και φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να είναι από την εποχή του Ρωμαϊκού Δικαίου. Αλλά πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να έχει μέλλον. Πιέζεται προς την κατεύθυνση αυτή. υπάρχει το θέμα του μονοπωλίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πολύ ωραία το εξηγήσατε ότι υπάρχει μια μικρή γκρίζα ζώνη αλλά αρκετά μεγάλη για να δράσει κανείς, είναι κάπως σκούρο γκρι. Και το γεγονός, τι θα πει καλή, ε, καλή, παρακαλή, σας παρακαλώ μήπως μπορείτε να κάνετε τίποτα, invite είναι αυτό στα αγγλικά, μήπως να έχουμε μια πιο έντονη διατύπωση γιατί ε, θα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δράσει. Επειδή έχω εργαστεί σε αυτά τα θέματα πολύ, όχι μόνο σε αυτή τη θητεία και σε κάποιο βαθμό στην περασμένη θητεία, έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τρελαίνεται κιόλα να επιτύχει αυτό το εργαλείο παρόλο που διαρριγνύει τα ημάτια τη, ότι βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο κοντά στους πολίτες. Εγώ βλέπω μια αντίφαση έτσι σε αυτό. Πώς τα βλέπετε παρακαλώ αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και εμά. Ενδιαφέρουσα ερώτηση πραγματικά. Ας σταματήσουμε εδώ και να σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε οι τρεις σας ε, στις δύο ερωτήσεις των εισηγητών και μετά θα δώσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε? Ωραία. Ο κύριε Σντεχρότ. Μπορώ να αρχίσω εγώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει ε, με το παραδεκτό και το άλλο ε, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο δεδειγμένος φορέας για να κάνει αυτό τον έλεγχο. Όπως είπε ο James Όργαν, ε, είναι νομικός έλεγχος αμυγός και σε τελική φάση όμως αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την πολιτική παρακολούθηση συνέχεια που μπορεί να μας ικανοποιεί ή να μην μας ικανοποιεί. Μπορεί ε, νομικά ε, ε, αυτό να επιτρέπεται, αλλά πολιτικά δεν είναι και πάρα πολύ επιθυμητό αν υπάρχει πολιτική σύγκρουση συμφερόντων δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί, αλλά ευσταθεί το επιχείρημα. Από την άλλη, ταυτόχρονα εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι υπάρχει και δικαστική ε, επίβλεψη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο στάδιο του παραδεκτού και του ελέγχου του κατά πόσο είναι παραδεκτή μία πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη νυν επιτροπή ε, το μόνο που έχει απορρίψει ως πρωτοβουλία ήταν το Stop Brexit. και θα σας πρότεινα να το σκεφτείτε κι εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή ληφθεί η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς τι κάνετε. Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα τόσοι Ευρωπαίοι πολίτες και τα πράγματα τελειώνουν εκεί τις περισσότερες φορές. Ποιος είναι ο απότερος στόχος μας. Είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος κάποια πράγματα, είναι να ε, συμμετέχουν οι πολίτες, είναι να χαράξουν την πολιτική ατζέντα, να καθορίσουν ποια θέματα θα συζητούνται. Είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί είναι ενδιαφέρον για τους διοργανωτές και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ε, να τα δουν αυτά για να επενδύσουν. Πολλές φορές δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους και για να μπορέσει να ευδοκιμήσει μία ε, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και να πιάσει και τόπο, θα πρέπει να ξέρουμε σε τι αποσκοπεί. Είδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είστε πραγματικά ε, μια βουλή εκπροσώπων από διάφορα κράτη-μέλη και γίνεται μια υπερεθνική συζήτηση, ε, νομίζω ότι εδώ θα βοηθήσει να ασχοληθείτε με αυτό. Αυτά. Και με χαρά να συζητήσουμε και περισσότερο για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, να το θέσω έτσι. Συμφωνώ με τον Μάρτιν ότι στο παρελθόν είδαμε και το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Και μπορεί να αποφασίζει να ανατρέψει ένα αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κατάλληλο θεσμικό όργανο να, για να ελέγξει κατά πόσον πρέπει να καταχωρηθεί μια πρωτοβουλία πολιτών ή όχι. Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδο αυτή τη μερική καταχώρηση, διότι στην αρχή οι πρωτοβουλίε των πολιτών απλώς αγνοούνται γιατί υπήρχαν ένα-δυο σημεία στην πρόταση που δεν ήταν σωστά βάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω όμω ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση και ε, υπάρχει πλήρης υποστήριξη για μερική καταχώρηση και από εκεί και πέρα μπορεί να εξηγήσουν στους πολίτες γιατί ε, δεν γίνονται δεκτά κάποια σημεία ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και να καταχωριστούν και αυτά τα σημεία. Και επίσης να πω ότι η διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα την οποία προετοιμάζουμε θα έχει και ένα help desk για τις νομικές συμβουλές. Αυτές οι νομικές συμβουλές δεν ε, θα είναι αμυγό επίσημε συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται λοιπόν για συμβουλές τι οποίε θα δίνουμε εμείς, η ΙΚΑΣ, σε συνεργασία με νομικού εμπειρογνώμονε στην Ευρώπη. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν γίνει κάποια βήματα ε, ώστε να συνεργαστούμε εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσουμε τους διοργανωτές των πρωτοβουλειών να καταχωρήσουν τις προτάσεις τους. Ίσως λοιπόν αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα, να μην ε, κρίνει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και κάποιοι άλλοι τρίτοι που ασχολούνται στην, με το ίδιο θέμα. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάτι το οποίο ευαισθητοποιεί τους πολίτες και μπορεί να είναι ένα μέσο που έχουμε στη δημόσια ε, σφαίρα. Είναι το μόνο διασυνοριακό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο ε, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πολιτών σε διάφορα κράτη-μέλη για να κινηθούν προς ένα ευρωπαϊκό στόχο. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές επικρίσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Αλλά όταν εμεί υποστηρίζουμε διοργανωτέ των πρωτοβουλειών, του λέμε σαφέστατα τι μπορούν να πετύχουν και τι δεν μπορούν. Πολλέ φορέ η απάντηση που λαμβάνουμε είναι ναι το ξέρω, θέλουμε ακόμα να την προωθήσουμε γιατί τη χρησιμοποιούμε ω εργαλείο ώστε ε, να μαθευτεί το θέμα το οποίο μα ενδιαφέρει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν οργανώσει και πολίτε που χρησιμοποιούν την πρωτοβουλία πολιτών για να διαβάσουν ένα μήνυμα. Και αυτή είναι μια σημαντική πτυχή. Και το τρίτο, για την ε, πρόσκληση προς την Επιτροπή, το κάλεσμα προς την Επιτροπή. Φυσικά και εν τέλει τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά δεν είναι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη και τους πολιτικούς εν γέννη. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση και να δείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αιρετοί ευρωβουλευτές μπορούν πραγματικά ε, να κάνουν κάτι για το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Ναι, φυσικά η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ουσιαστική εδώ. Η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ασυνήθιστος φορέας. Έχει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και διστάζω να πω ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού, αλλά είναι πολύ ασυνήθιστο. Και όσον αφορά το θέμα της καταχώρησης, για το κατά πόσον κρίνουν και αποφασίζουν οι ίδιοι, ε, έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα το διαχειριστεί κάποιος και αν θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό. Από την υπόθεση του TTIP και μετά, εμπλοκή του δικαστηρίου ήταν αυτό το οποίο έλυσε τελικά την διαμάχη στην ε, ε, υπόθεση της ε, TTIP. Βέβαια η ταχύτητα της απάντησης σε ένα ερώτημα είναι θέμα για τους διοργανωτές των πρωτοβουλειών και φυσικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μετά από την δικαστική απόφαση. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του ενδιαφέροντος θα πρέπει να παραμείνει αλλά η σύγκρουση συμφερόντων αλλά εάν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να άρουμε τη σύγκρουση συμφερόντων τότε καλό, καλύτερα θα ήταν. Ε, πολλοί χρησιμοποιούν όντω την ε, πρωτοβουλία πολιτών για κινητοποίηση και εκστρατεία και φυσικά η συνέχεια που θα δοθεί ε, πρέπει να απηχεί ακριβώ και τη φωνή ε, των πολιτών των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι επιπλέον για το στάδιο της συνέχειας υπάρχει ένα κενό ως προς τις προδοκίε, και αυτό που θα μπορούσε ίσω να κάνει με, η μεταρρύθμιση είναι ότι προφανώς υπάρχουν διοργανωτέ που θέλουν τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις δικές τη διαδικασίες πολιτική και ακολουθούν τις ε, διαδικασίες τους. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό μεταξύ αυτών που περιμένουν οι διοργανωτέ τη πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι εφικτό. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί ότι απαντά και οι διοργανωτέ τη πρωτοβουλία να μην είναι ικανοποιημένοι και να λένε ότι συλλέξαμε ένα εκατομμύριο υπογραφέ και η Κομισιόν αδρανεί. Νομίζω λοιπόν ότι στην όλη διαδικασία τη συνέχεια κάποια από τα εργαλεία και οι ιδέε που χρησιμοποιήσαμε είναι ακριβώ για να κλείσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει και να μπορέσουν να συμμετέχουν και πολίτε ε, και σε ακροά στο και σε συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία πολιτών, για να μειώσουμε το χάσμα και να βελτιώσουμε και τη χάραξη τη πολιτικής. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που μας παρουσίασαν τις απόψεις τους και θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα θέματα και να υποβάλω και κάποιες ερωτήσεις. Εκείνο που με ανησυχεί είναι η κατάσταση υγείας της Ευρωπαϊκής ε, Πρωτοβουλίας Πολιτών. Δηλαδή, να εξηγηθώ, βρίσκεται πολύ κοντά σε αρρώστια το ECI και υπάρχει κίνδυνος ε, αυτή η πρωτοβουλία να καταστεί ένα παιχνίδι κυρίως στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δοθεί εντύπωση στους ε, πολίτες ε, ότι δήθεν συμμετέχουν αλλά κατ' ουσίαν να τους απαγορεύουν να συμμετέχουν στις πολιτικές που χαράσουν οι θεσμοί ή τα κράτη-μέλη. Αυτός λοιπόν ο κίνδυνος για μένα είναι πολύ μεγάλος και εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Με ποιον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να μετατραπεί σε κάτι ε, πολύ πιο εξελιγμένο και πολύ πιο δαπανηρό από τις απλές αναφορές. Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους ε, πολίτες. Αν όμως πραγματικά θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά το παιχνίδι αυτό και το να το μετατρέψουμε σε ένα όπλο στα χέρια των πολιτών, κατά την άποψή μου τότε θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα ε, τα οποία θα έχουν και σχέση με τις επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν τα σοβαρά μέτρα είναι πρώτα απ' όλα να περιορίσουμε τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις ε, φάσεις ε, δημιουργίας του ECI από το επιτρεπτό ε, στην ε, καταχώρηση και στο follow-up. Να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων και να αναθέσουμε σε μια τρίτη αρχή την ε, δυνατότητα να κρίνει την, το αρχικά παραδεκτό, την έγκριση, την αρχική έγκριση της πρωτοβουλίας. Ε, δεν ξέρω ποιος την έκανε αυτή την πρόταση, νομίζω ο πρώτος ε, ομιλητής, θα πρέπει να εξηγηθεί ποια θα πρέπει να είναι αυτή η τρίτη αρχή. Εγώ σκέφτηκα τον ε, διαμεσολαβητή, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Και να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτή την τρίτη αρχή με τις αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεύτερο σημαντικό μέτρο θα ήταν μια ευρεία ερμηνεία του πεδίου ε, αρμοδιοτήτων και εφαρμογής του ECI, κυρίως όσον αφορά την αναδιατύπωση της ε, νομικής πράξης, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ε, τα, οι προκατακτικές πράξεις που προηγούνται των νομοθετικών πράξεων. Να υπάρχει δυνατότητα, αναφέρθηκε, να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Αυτές είναι αυτό σημαίνει αλλαγή, τροποποίηση των συνθήκων έτσι ώστε οι συνθήκες ε, να εμφανίζονται ως μέτρα για να βελτιώνονται οι ίδιες οι συνθήκες, κυρίως με αναφορά στο άρθρο υπαριθμών 3. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, αρκετά ενδιαφέρον, όπως το ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Όργαν, ε, να γνωρίζουμε δηλαδή με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει νόμιμα διάφορα στοιχεία της συνθήκης ε, για να είναι δυνατόν να λάβουν χώρα αυτές οι τροποποιήσεις. Ε, προφανώς η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της άρνησης, αλλά τελικά αν απευθυνθούμε σε μια τρίτη αρχή για να παρεμβαίνει εκείνη στην ε, φάση της ε, καταχώρησης, δεν θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο διαμεσολαβητή. Και τέλος, η μερική καταχώρηση που περιλαμβάνεται στη νέα πρόταση της Επιτροπής. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν είναι αυτό εκείνο το οποίο θα μετατρέψει το ECI σε κάτι διαφορετικό από παιχνίδι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Μπάρμπαρα. Πραγματικά απολαμβάνω πάντα να σας ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, είμαστε λίγο υποπίεση χρόνου. Και ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ε, παρακαλώ. Ο κύριο Τερικάμπρα, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, γιατί με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Και εγώ τα έχω επαναλάβει πολλές φορές, αλλά έχω τέσσερα σημεία που είναι τόσο σημαντικά που είμαι υποχρεωμένος να τα ξαναπώ. Τι να κάνω. Η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν θα αναφέρω. Να πω τέσσερα άλλα πράγματα. Εξ ονόματος ε, της ομάδας των Πρασίνων Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, το πεδίο εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περιοριστική διατύπωση, πολύ στενή. Εμείς θέλουμε να συμπεριληφθούν και όλες οι πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών που ε, από τον ένα θέματος ενός θέματος ε, για το οποίο έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθετική ε, πράξη, την κατάργηση, τροποποίηση, αναδιατύπωση οποιασδήποτε πράξης. Δεύτερον, επανειλημμένα ακούστηκε και προτείνουμε και εμείς να συσταθεί ένα ανεξάρτητο σώμα και δεν το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει τον έλεγχο του παραδεκτού. Τρίτον, συνέχεια η παρακολούθηση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει τίποτα καινούριο. Η ομάδα μας περιμένει εξορισμού πρόταση για νομική πράξη και ενίσχυση της διατύπωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να τεκμηριώνει απολύτως και πλήρως και λεπτομερώς την ε, αντίρρηση και την άρνηση να προβεί σε δράση. Και τέταρτο και τελευταίο, ε, συνέχεια που πρέπει να δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτε εδώ προτείνονται αλλαγέ. Εμεί προτείνουμε συζήτηση στην Ολομέλεια με ψηφοφορία και ψήφισμα με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν χρειάζεται να ε, προτείνει νομική πράξη συν τη δυνατότητα να προτείνει έκθεση ε, ιδίας νομοθετικής πρωτοβουλίας σε περίπτωση που δεν αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τερή Κάμπρας γρήγορα να απαντήσουμε και σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Κύριος Δεχρότ. Um, I think that... Νομίζω ότι ήταν μάλλον δηλώσεις και λιγότερο ερωτήσεις. Θα απαντήσω σύντομα σε αυτά που ανέφερε η κυρία Σπινέλη. Δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να καταντήσει αναφορά. Υπάρχει αναφορά. Ε, πώς θα διατηρήσουμε το υψηλό προφίλ και την υψηλή αξία. Ε, για να έχει νόημα θα πρέπει να ε, δοθεί αξιόπιστη συνέχεια στις υφιστάμενες παραδεκτές ε, πρωτοβουλίες. Μέχρι στιγμής ε, λαμβάνουν γραπτή απάντηση και κλεισμένο των θυρών συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ε, ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα τι. Δεν αρκεί αυτό. Άλλη μια δημόσια ακρόαση ενέφερα εγώ ε, ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γενικότερα εμείς πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο υπάρχει για να δίνει συνέχεια στη συζήτηση και με τους διοργανωτές που θα πρέπει με διαρθρωμένο τρόπο να συμμετέχουν στο διάλογο και να τονίσω κάτι που ακούμε πολύ ότι Καλά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει δημόσιες ακροάσεις έτσι κι αλλιώς. Την έχει αυτή την εξουσία ή να κατεβάσει ψηφίσματα. Αλλά δεν είναι τυποποιημένη αυτή η διαδικασία στάνταρ. Βέβαια, να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν θα γίνει ψηφοφορία ή όχι για μια πρωτοβουλία. Όχι, να τυποποιηθεί, να κατοχυρωθεί και να είναι στάνταρ διαδικασία για όλες τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες. Η κυρία Λιρώνη, ε, θα συνοψίσω λίγο απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. Ένα φόβο έχω εγώ. Ε, για το θέμα του παραδεκτού αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προχωρεί στην καταχώρηση ε, των πρωτοβουλειών και δεν δίνει συνέχεια με κάτι συγκεκριμένο, ε, υπάρχει κίνδυνος ότι αν το αναθέσουμε αυτό σε ένα τρίτο φορέα, χαιρετίσματα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που η ίδια αυτή τη στιγμή τα δεν τα συνεχίζει. Τώρα άμα το αναλάβει ένας τρίτος, ε, δεν πρόκειται να αντιδράσει. Ακόμα πιο δύσκολο ας πούμε. Και δεν θα το συνιστούσα. Πάντως επιμένω ε, στην επιγραμμική πλατφόρμα ε, συνεργασίας ε, με προτάσεις κτλ. Αυτό όμως είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, θα δούμε πώς θα πάει. Και γενικά θέλω να πω κάτι. Εκπλήσωμαι πάρα πολύ που ακούω τόσους ευρωβουλευτές να λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν λειτουργεί. ακόμα θεωρείται έτσι παιχνιδάκι, ενώ εμείς που είμαστε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πραγματικά συμφωνούμε και μην περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας αποδείξει ότι είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Κάντε εσείς στο Κοινοβούλιο. Δείξτε ότι είστε πρόθυμοι να δεχτείτε τη συμμετοχική ε, δημοκρατία. Οι πολίτες εσάς ψήφισαν, εσάς εξέλεξαν, όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς τους εκπροσωπείτε. Χαίρομαι να ακούω που λέτε ότι το ECI είναι παιχνιδάκι αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα σας να πείτε και να δείξετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παίρνει σοβαρά υπόψη τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών να το φέρτε στην Ολομέλεια να το ψηφίζετε και να δείξετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, κανείς δεν σας υποχρώνει να υπερψηφίσετε μια πρωτοβουλία πολιτών με ένα εκατομμύριο υπογραφέ, μπορείτε κάλλιστα να την καταψηφίσετε. Αν θέλετε να πείτε ότι είναι σοβαρό και δεν είναι παιχνίδι, κάντε το. Τώρα εγώ πώς να συνεχίσω μετά από όλα αυτά. Ε, μερικά σχόλια, λέει κύριο Σόργαν, για το θέμα των εξαρτήτου φορέα. Υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προάγει την ε, δημοκρατία και έχει νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιεί στο μέλλον, το άρθρο 11 κτλ. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία πολιτών. Μετά από 20-30 χρόνια μπορεί να υπάρχουν άλλα εργαλεία που θα χρειάζονται ανεξάρτητο οργανισμό για να διαχειριστεί αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Ε, μ' άρεσε αυτό που είπε η κυρία Σπινέλη για την τροποποίηση των συνθηκών, είναι σημαντικό. Στι προπαρασκευαστικέ δράσει δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτική διαδικασία και το Συμβούλιο τελικά μπορεί να τα απορρίπτει. Και συμφωνώ με την ε, Ελίζα, είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου να κινήσει διαδικασίε. Σα ευχαριστώ όλου που αποτελήσατε πηγή έμπνευση και επαφήθηκε την, ε, στην εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου όλο αυτό το θέμα. Να δώσω τώρα το λόγο στην Τανούτα Χούμπνερ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων και θα σας δώσω συμβολικά ε, τα ενία για να προεδρεύσετε στο δεύτερο ε, τμήμα ε, της ακρόασης. Είναι πολύ πειθαρχημένο το κοινό και δεν θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι, απλώς ε, να σας καλωσορίσω όλους και εγώ με τη σειρά μου και να σας πω ότι τώρα περνάμε στο δεύτερο πάνελ και το δεύτερο πάνελ αυτής τη ακρόαση αφορά την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς από αυτούς τους ανθρώπους που αποκαλούμε practitioners ε, στην ε, ορολογία των Βρυξενών, όλους αυτούς που καταπιάνονται με τα θέματα αυτά ε, και θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο από την ευρωπαϊκή αλλά και από τις εθνικές εμπειρίες και θα πρέπει να μάθουμε όχι μόνο από τα αποτυχημένα παραδείγματα, αυτά τα οποία δεν μας οδήγησαν σε τίποτα, αλλά και από τα επιτυχημένα παραδείγματα. Περιμένουμε λοιπόν κάποιες σημαντικές πληροφορίες από το δεύτερο πάνελ για μας ως νομοθέτες και επίσης θα ήθελα να σας πω διότι από την πρώτη στιγμή και Τζόρτζ μιλώ λίγο εκ μέρου σου ε, από τότε που αναλάβαμε εμείς ε, εδώ αυτή τη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με την πρωτοβουλία πολιτών γιατί όλοι δεσμευόμαστε ε, να έχουμε αυτή την Ευρώπη η οποία θα ξεκινά από τη βάση προς την κορυφή και να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες στη διαμόρφωση της Ευρώπης και αυτό σημαίνει διάλογος με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επίσης εξετάζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών και την πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού ε, εδώ και ε, κάποιο διάστημα για την τελευταία χρονιά. Η πρώτη πρόταση του George Σέπφιλ ήταν το 2015 και Συζητούσαμε και με τον Φραν Τίμερμαν, ο οποίο και αυτό ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και ε, μοιραζόμαστε μαζί του ιδέε που ε, μα δίνετε κι εσεί ε, και έχουμε και την εμπειρία των θεμάτων αυτών και επομένω σήμερα δεν έχουμε μόνο την εμπειρία των συζητήσεων και αυτά που γνωρίζουμε από εσά, από του ανθρώπου που ασχολούνται με το θέμα αυτό και είναι εμπειρογνώμονε, αλλά υπάρχει και σημαντική νομολογία που νομίζω ότι είναι επίση ε, σημαντικό, διότι διευκρινίζει και τα καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τα, η καταχώρηση των ετοιμάτων και δίνει και κάποιε διευκρινήσει για τη φύση των πρωτοβουλειών που μπορούν να καταχωριστούν και ε, ένα βαθμό σε έναν βαθμό και μια αιτιολόγηση που χρειάζεται για τις αποφάσεις. Επίσης ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ήδη το σχέδιο έκθεσης και ο Τζόρτς κάποια στιγμή θα αναφερθεί σε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ε, έχουμε ε, τη συνεδρία τη Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων που θα συζητηθεί αυτή η έκθεση. Θα ψηφίσουμε και θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια και ελπίζουμε στο μεταξύ ε, να τροποποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, γίνει μια καλύτερη πρόταση χάρη σε εμά. Να δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές μας. Από τη Λετωνία έχουμε τον κύριο Ήμαρτς Πράιταξ. Στη συνέχεια από το Right to Water, ε, την πρωτοβουλία αυτή, τον Βίλεμ Γκούντριαν και τον κύριο Μπάλας Τάρνοκ από την Ένωση Ράκοτσι από την Ουγγαρία να δώσω πρώτα το λόγο στον Ήμαντς Μπράινταξ να μας κάνει την παρουσίασή του. Ε, οι κανόνες είναι οι ίδιοι για ο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι καλό να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και ελπίζουμε ότι κάποια από τα πράγματα που καταφέραμε σε εθνικό επίπεδο θα μπορέσουν σε κάποιο βαθμό να ε, χρησιμοποιηθούν και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ο στόχος μου εδώ σήμερα είναι με δύο λόγια να εξηγήσω τι είμαστε, τι κάνουμε και πώς γίνεται αυτό. Και μετά να σας παρουσιάσω και κάποια συμπεράσματα για το πώς θα μπορούσε να ε, γίνει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γιατί είχε αποτέλεσμα στη Λετωνία. Η Maribals.lv είναι μια ε, πρωτοβουλία πολιτών στο διαδίκτυο, ε, πλέον γίνεται τεσσάρων ετών και είναι μια πλατφόρμα στην οποία οποιοδήποτε πολίτης ε, στη Λετωνία από 16 ετών και πάνω μπορεί να υποβάλει μία πρόταση. Αυτά δεν είναι πλήρη νομικά κείμενα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι κανεί ε, νομικό. Ε, πρέπει να έχει σώσει τα βέβαια, αλλά αυτό δεν είναι τη παρούση. Δεν χρειάζεται όμω να είναι κάποιο νομικό για να γράψει. Εμεί κάνουμε έναν έλεγχο ποιότητα αυτού που υποβάλλεται και ε, δημοσιεύουμε τι θέλουν οι πολίτες. Δεν γράφουμε το κείμενο, αλλά σχολιάζουμε και προσπαθούμε να προσφέρουμε και κάποια υποστήριξη. Αυτό είναι αποτελεσματικός τρόπος ε, ε, με τον οποίο εδώ και 7 χρόνια οι πολίτες στη Λετωνία επηρεάζουν και έχουν αλλάξει και νομοθεσία. Είναι ένας μηχανισμός ψηφιακής επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν αφορά μόνο τους διάφορες παράγοντες και όλους εκείνους που θα βρουν έναν τρόπο να επηρεάσουν τα πράγματα. Ε, θα βρούνε ε, τον δρόμο ακόμα και μέσω της πιο περίπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας. Αυτό είναι για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο, που έχουν κουραστεί ε, να ψηφίζουν ε, για αμφισβητούμενα ζητήματα και έχουν κουραστεί από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και θέλουν να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε, θέλουμε να έχουμε όλο και περισσότερους και μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει. Όσον αφορά τα ποσοστά επιτυχίας, το 50% των πρωτοβουλίων των πολιτών που ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο από την πλατφόρμα μας ε, ε, εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο ή σχεδόν εγκρίθηκαν. Θεωρούμε ότι επιτυχές ε, αποτέλεσμα ακόμα και μια ε, μερική νίκη. Ακόμα και αυτή τη θεωρούμε νίκη. Και αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 17 ή 18 αλλαγές στην νομοθεσία μέχρι τώρα. Δεν είναι τεράστιος ο αριθμός όσον αφορά το νομοθετικό έργο, αλλά αν δούμε τα στοιχεία συνολικά, υπάρχουν ε, στοιχεία που δείχνουν ότι είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, διότι 70% των πολιτών έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα τουλάχιστον μία φορά. Και Βέβαια, όλοι οι επισκέπτες ε, δεν ψηφίζουν απαραίτητο. Ε, αυτοί που ψηφίζουν είναι 220.000 άνθρωποι, είναι το 15% του εκλογικού σώματος και εξ όσων γνωρίζουμε είναι και ο υψηλότερος ε, αριθμός στον κόσμο αυτός. Και κάτι το ασυνήθιστο είναι ότι είμαστε και αυτάρκες από οικονομική σκοπιά, διότι μέχρι τώρα 28.000 άνθρωποι μας έχουν κάνει κάποιες μικροδωρεές. αν δίνει κάποιος 5.000 ευρώ σε ένα πολιτικό κόμμα, ε, σε εμά θα δώσει, όχι βέβαια ο ίδιος άνθρωπος, 2 ευρώ, 5 ευρώ ε, και στη δημοκρατία ούτως ή άλλως ε, δεν θα πρέπει να είναι η αγοραστική αξία κάποιου που μετράει, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Και φυσικά ε, χαιρόμαστε που αυτοί οι άνθρωποι μας υποστηρίζουν και οικονομικά. Αυτό μας επιτρέπει να επιβιώνουμε και μάλιστα γινόμαστε και πιο ισχυροί, καταφέρνουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή και καλύτερα αποτελέσματα κάθε χρόνο. 220.000 άνθρωποι λοιπόν έχουν ψηφίσει έστω μία φορά. Οι συνολικές ψήφοι είναι 950.000 ε, σε 2 ε, εκατομμύρια πολίτες. Ο μηχανισμός δουλεύει ω εξής. Γράφουν τις ιδέε οι πολίτες, τις στέλνουν σε εμά, ε, κάνουμε έναν ποιοτικό έλεγχο, τι δημοσιεύουμε και από εκεί και πέρα ξεκινά η ψηφοφορία. Όταν ε, συλλεχθούν 10.000 υπογραφές, ε, βάσει τη νομικής διαδικασίας το Κοινοβούλιο πρέπει να το αναθεωρήσει, να το εξετάσει το ζήτημα και να ψηφίσει. Και μάλιστα το Κοινοβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις ε, ανέλαβε πρωτοβουλία ακόμα και με χίλιες ή δύο χιλιάδες ή τρεις χιλιάδες ψήφους εάν κάποιος στο Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι ένα φλέγον θέμα σε πολιτικό επίπεδο, τότε το λαμβάνουν υπόψη. Διότι 10.000 υπογραφέ είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, ε, γιατί είναι περίπου το 0,5% του πληθυσμού και είναι πολύ μεγάλος ε, αριθμός αυτός. Όταν όμω φτάσουμε στις 10.000 υπογραφές, ε, είναι λίγο δύσκολο να γνωρίσει κανεί αυτή την εντολή. μα λυπεί βέβαια οποιαδήποτε απόρριψη, αλλά ε, αν συνολικά έχουμε ένα επιτυχημένο ποσοστό, τότε δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα. Τώρα, πώς λειτουργεί σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες αντίστοιχες ε, και γιατί η Λετωνία έχει κάνει κάτι ε, το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε, το 90% αντίστοιχων πρωτοβολιών δεν έχουν καταφέρει και δεν υπάρχει κάτι σε αντίστοιχη πλατφόρμα. Καταρχάς αυτές είναι νομικές ιδέες, δεν είναι πλήρη νομικά κείμενα και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται αυτομάτως ο αριθμός των πολιτών που μπορούν να ε, ε, συμμετέχουν. Χρησιμοποιούμε ε, εργαλεία έγκρισης, τα οποία σημαίνει ότι οι πολιτικοί δύσκολα μπορούν να τα αγνοήσουν. Αυτά γίνεται με ψηφιακές τράπεζες και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος πολιτικός ο οποίος θα αμφισβητήσει σοβαρά τον αριθμό των υπογραφών. Ε, Υπάρχουν επίσης κάποιες περιπτώσεις και νομίζω ότι εδώ ε, μπορώ να πω ότι η Φιλανδία Ε, έχει το εξή. Ε, η αντιπολίτευση ουσιαστικά έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των πολιτών, που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον μια πρωτοβουλία των πολιτών, αλλά είναι ένα κίνημα ενό πολιτικού κόμματο. Έχουμε και εμεί κάτι αντίστοιχο από πολιτικά κόμματα, αλλά έχουμε καταφέρει να τα περιορίσουμε με επιτυχία. Και αν ε, δούμε το πώς λειτουργεί σήμερα και πώς λειτουργεί η πρωτοβουλία πολιτών, εμείς ε, ε, έχουμε ως κινητήριο μοχλό την ανάγκη ουσιαστικά. Βοηθούμε τον κάθε πολίτη να τα διαμορφώσει με τρόπο ώστε να μπορεί να περάσει στα μέσα. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί όπως προς τα μέσα για το χώρο ε, στην αγορά. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο ισχυροί με τα μέσα, αλλά βοηθούμε να διαμορφωθεί το μήνυμα κατά τρόπον ώστε να είναι ενδιαφέρον και να επιθυμούν και οι πολιτικοί να εμπλακούν. Ε, δίνουμε δηλαδή ουσιαστικά στους πολίτες τις ιδέες ε, σε δημόσιες σχέσεις που αγοράζουν οι περισσότεροι με χρήματα και εμείς τις προσφέρουμε στους πολίτες δωρεάν. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους πολύ δύσκολα μπορούμε να δώσουμε τεχνογνωσία στους υπολείπους, διότι παραδοσιακά ε, οι απλοί πολίτες δεν καταφέρνουν πολύ εύκολα να ε, κάνουν εθνικές εκστρατείες ε, χωρίς χρήματα και η ε, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είναι τόσο δαπανηρή που δεν έχει κανείς την οικονομική δυνατότητα να τους προσλάβει. Περνάει η ώρα βέβαια. Να σας πω λοιπόν πώς μπορούμε να περάσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών από μία απλή απόδειξη ότι υπάρχει μια ιδέα σε, ε, να γίνει ένα λειτουργικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας. Ε, υπάρχουν ακτιβιστές βέβαια που είναι πάρα πολύ δραστήριοι και καταφέρνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ε, κατά μέσο όρο οι πολίτες... Ε, έχουν ουσιαστικά τρία λεπτά στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν την άποψή τους και πρέπει να είναι κατανοητό το μήνυμά τους, πρέπει να είναι ισχυρό αλλά εύκολο αυτό που προσπαθούν να κάνουν και η υπερβολική γραφειοκρατία και η υπερβολική διαχείριση στη δημοκρατία δεν θα βοηθήσει. Το σύστημα ελέγχου της ποιότητας ε, ε, είναι αυτό το οποίο μας βοηθά. Δημοσιεύουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που λαμβάνουμε. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμωμένοι, μας λένε ότι είμαστε πράκτορες της Washington, δεν μας λένε ότι είμαστε Κινέζοι βέβαια, οπότε καλό είναι και αυτό. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία φυσικά δεν θα δημοσιεύσουμε ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών ε, να αναθεωρήσουμε και την δυνατότητα επιρροής που υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιον απευθύνουμε τις πρωτοβουλίες και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα πρέπει να ε, προχωρήσει από το εθνικό επίπεδο και πάνε. Δεν υπάρχει ενωμένος χώρος, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται σε εθνικό επίπεδο υπάρχει πολωνικός χώρος ε, πληροφοριών, ισπανικός, ε, λετονικός και υπάρχει αλληλεπίδραση μόνο σε μερικά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να υπάρχει εθνική παρουσία και μετά πέραν αυτού μπορεί να έρθει να προσθέσει και ένα 5% ευρωπαϊκών θεμάτων. Ε, δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τους πολίτες να εγκρίνουν ευρύτατα ένα θέμα αν δεν υπάρχει εθνική παρουσία για το θέμα. Γι' αυτό ακριβώ και θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε την εμπειρία μας σε άλλες χώρες, αλλά πρώτα σε εθνική κλίμακα. Ε, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα, Συμβούλιο της Ευρώπης και εθνικά ε, θεσμικά όργανα, είπαμε πρέπει να συμμετέχουν. Ε, σε 10 ε, χώρες μία λειτουργική εθνική πλατφόρμα αρκεί θεωρούμε για να μπορέσουμε στη συνέχεια να έρθουμε να προσθέσουμε και το ευρωπαϊκό επίπεδο και ο αριθμός των υπογραφών θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να είναι 2,5 εκατομμύρια διότι κάνουμε μια προβολή σε σχέση με τη λετωνική εμπειρία. 10.000 ε, υπογραφέ είναι το 0,5%, επομένω σε ευρωπαϊκού όρου θα πρέπει να είναι 2,5 εκατομμύρια. Αλλά φανταστείτε ποια θα είναι η εντολή για μεταρρυθμίσεις, για προτάσεις, εάν για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσει να ε, έχει μια νέα ιδέα ε, για κοινό στρατηγείο για τις ευρωπαϊκές χώρες ε, και υπάρχουν 20 εκατομμύρια υπογραφές για το θέμα αυτό. Η εντολή είναι πολύ πιο ισχυρή. Έχω την εξή ερώτηση. Υπάρχει ψηφιακό μάρκετινγκ στην περιοχή στην οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα και αν υπάρχουν ε, νομοθετικοί φορεί οι οποίοι ε, σέβονται και την πίεση λόγω του αριθμού υπογραφών για μία πρόταση. Αν η απάντηση είναι κατευθυντική και στα δύο, τότε η εμπειρία τη Λετωνία αποδεικνύει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν απαιτεί 5 ή 50 χρόνια για να περάσουμε από όλε τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε για να τα καταφέρουμε. Η εμπορία της Λετωνίας δεν είναι θεωρητική, είναι πρακτική και ε, μπορούμε να σας αποδείξουμε πώς μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και επίσημα στοιχεία και επίσημοι φορείς, αλλά ε, δεν ξεκινά έτσι μια δέσμευση. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική βούληση και αυτό περιμένω να δω όλο και περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που μου επιτρέπετε να είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι αντιπρόεδρος ε, της ε, πρώτης επιτυχημένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και ε, Γενικός Γραμματέας ε, της Μονάδας ε, Δημόσιων Υπηρεσιών που είναι και η κινητήρια δύναμη πίσω από όλο αυτό. Να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές αλλά και τους ακτιβιστές, αυτούς που οργάνωσαν την εκστρατεία που μας βοήθησαν να στήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Επίσης είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που έχουμε επιτύχει και ελπίζω πολλοί που βρίσκεστε στην αίθουσα να έχετε υπογράψει για αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή συγκρίνεται και με την οδηγία περί πόσιμου ύδατος ε, που ίσως έχετε δει ε, φωτογραφίες. Ο κύριος ε, Τίμερμανς ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι μετά από πέντε χρόνια ανταποκρίνεται σε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, λίγη ιστορία για αυτή την ε, πρωτοβουλία. Ε, πολλοί ξεχνάνε ότι είναι μια πρωτοβουλία που ε, προέκυψε μέσα από αγώνες εθνικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το νερό, έτσι ώστε το νερό να παραμείνει σε δημόσιους οργανισμούς το νερό είναι δημόσιο αγαθό και το βασικό μας αίτημα ήταν να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία όπου ε, θα αναγνωρίζεται το πόσιμο είδωρο ως ένα δικαίωμα όπως το αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, η οδηγία περί πόσιμου ύδατος ε, ανταποκρίνεται εν μέρη αλλά όχι πλήρως. Επίσης, καλούμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ε, κάτοικοι θα έχουν δικαίωμα σε πόσιμο είδωρ. Ε, επίσης, ε, τα σώματα υπέρ της διαχείρισης των υδάτιων πόρων, αυτοί να μην υπάγονται στους κανόνες της αγοράς, να αποκλείονται από την απελευθέρωση και ε, η επιτυχία που υπάρχει είναι ότι οι υπηρεσίες συντάτων δεν εντάσσονται ε, στην εσωτερική αγορά. Και υπήρχε και ένα αίτημα να ε, ενταθούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει γενικώ και παγκόσμια πρόσβαση σε πόσιμο είδος και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Επιτυχημένη λοιπόν, επιτυχημένο το ιστορικό, έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Ε, καταρχήν, ένα κόμμα, περίπου 1,9 εκατομμύρια υπογραφές σε αυτή την πρωτοβουλία ε, ε, την, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ίσως κάποιοι από εσάς να θυμάστε ότι ο Επίτροπος Μπαρνέ απέκλεισε την οδηγία ε, περί δημοσίων ε, συμβάσεων ε, κατόπιν το 2013 υπήρχε η όλη συζήτηση γνωρίζουμε ότι όσοι δεν μπορούν να περάσουν και θέσει τους επανέρχονται και έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να προετοιμάζει τον δικό της τον αγώνα έτσι ώστε το όλο θέμα να επανέλθει σχετικά με τις οδηγίες. Μία άλλη επιτυχία αφορά τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Όπως σας είπα, ε, δεν ε, καταβάλλονται προσπάθειες απελευθέρωσης για το νερό. Και τέλος, να μην ξεχνάμε μεγάλη επιτυχία της πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο. Σε αρκετές χώρες, Σλοβενία, Έχουμε δει λοιπόν αρκετές χώρες ε, στην Ιρλανδία, εκεί είχαμε μια μεγάλη εκστρατεία όπου οι πολίτες εμπνεύστηκαν από ε, πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες, στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα οι πολίτες ε, και οι εργαζόμενοι έχουν εμπνευστεί έτσι ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να μην ιδιωτικοποιηθούν τα ύδατα. Ε, όλα αυτά τα θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν δύο προβλήματα που εντοπίσαμε, ίσως να υπάρχουν και πολλά άλλα, αλλά δύο θεωρούμε εμείς ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά ε, και αναφέρονται στην ε, ημερήσια διάταξη για να σχολιστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Το ένα αφορά στην συγκέντρωση, στη συλλογή υπογραφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταθέτει μια συγκεκριμένη πρόταση, αλλά υπάρχουν και αρκετές διαφορές στα κράτη-μέλη για το ποια δεδομένα πρέπει να υποβληθούν. Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, ε, εκεί δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Ε, σε άλλες χώρες ε, πρέπει κανείς να προσθέσει και κάποια άλλα στοιχεία, ας πούμε τον αριθμό του διαβατηρίου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι περίεργο και πραγματικά αυτό δυσχεραίνει τη συγκέντρωση υπογραφών σε αρκετές χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θίξει οι πολίτες. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι έλλειψη εμπιστοσύνης, όμως οι το θίγουν αυτό το θέμα. Σε αρκετές χώρες όπως τη Γερμανία είχαμε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές για αυτή την πρωτοβουλία. Οι ε, δημόσιες αρχές δεν έχουν ε, κανένα πρόβλημα στο να ελέγχουν τις υπογραφές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το λάβει σοβαρά υπόψη του, να επανεξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε και στο δεύτερο θέμα. Ε, όπως είπαμε και εγώ και πολλοί άλλοι που στηρίζουμε την εκστρατεία, ε, έχουμε όσο πιο μεγάλη είναι η δέσμευση για τους πολίτες να προσφέρουν στοιχεία, τόσο πιο δεσμευτική θα πρέπει να είναι και η όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια πρωτοβουλία ε, η οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το πλαίσιο των συζητήσεων ε, σε μεγάλο βαθμό λέω, γιατί ακόμα δεν έχουν προκύψει πολλά άλλα πράγματα. Οι πολιτικές προεκτάσεις ε, και πώς ε, θα οργανωθούν αυτές, αυτό είναι κάτι που κατά την άποψή μου πρέπει να το εξετάσουμε. Υπήρξαν αρκετές συζητήσεις σχετικά με την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως σας είπα, εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων με ένα άλλο καπέλο, σε έναν άλλο τομέα είχα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραδείγματος χάρη στις ε, συλλογικές συμβάσεις. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προσπαθήσει σταδιακά ε, να επεκτείνει το ρόλο της, της αξιολόγησης. Όσο περισσότερο μπορεί κανείς να περιορίσει την αυθαιρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο καλύτερα για όλους μας. Η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ε, δεν μπορεί κανείς αυτό να το θεωρεί δεδομένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ε, ε, θα ήταν ε, φιλική αν ε, υπήρχε κάτι που θα την ενοχλούσε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Και εμείς μετά από πέντε χρόνια τώρα βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι που εμείς το υποτιμήσαμε γιατί δεν σταματάει κάπου το ECI. Πρέπει κανείς να συνεχίσει με αυτή την πρωτοβουλία. Ήμασταν πολύ ευτυχείς για το ότι το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία ε, να ε, τοποθετηθεί στην πρωτοβουλία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, τουλάχιστον όσον αφορά στον κανονισμό. Πώς είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πιο σημαντικές πολιτικές ομάδες να ε, στηρίζονται με υπογραφές και να συμφωνούν για τους στόχους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κάνει τίποτα. Μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει. Όπως σας είπα θα συνεχίσουμε να μιλάμε με ευρωβουλευτές, με προσώπους της Επιτροπής, γιατί έχουμε ως ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων τη δομή να το κάνουμε αυτό. Και η ομιλία περί πόσιμου ύδατος είναι τουλάχιστον μια μερική απάντηση στη δουλειά που έχουμε ήδη κάνει. Για να ανακεφαλαιώσω, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην συνεχιζόμενη υποστήριξή του και όπως είπε και ένας από τους προλαλήσαντες, θα επανέλθουμε για να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να μεταφράσουμε το ECI ε, με περαιτέρω βήματα. Θα μιλήσουμε με εσά και τους ε, συναντέλφους σας. Και υπάρχουν δύο θέματα που εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Το ένα είναι η συγκέντρωση των υπογραφών και το δεύτερο είναι το θέμα της ε, πολιτικής βούλησης. Να το βελτιώσουμε αυτό εκεί όπου συμφωνεί η Πρωτοβουλία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να καταθέσει κάποιες προτάσεις για μελλοντική πρόοδο. Ευχαριστώ κύριε Χαοντριάν. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τάρνοκ από την Ουγγαρία. Είναι από την Ένωση Ρακώση. Θα το πω στα αγγλικά γιατί στα αγγλικά έχω το κείμενο. είναι συντονιστής της πρωτοβουλίας Minority Safe Pack. Είναι μια πρωτοβουλία που συλλέγει υπογραφές. Θυμάστε ίσως ότι στο Λουξεμβούργο προσέφηγαν κατά απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία ε, το 2013 ε, θέλησαν να την ε, υποβάλλουν. Το αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν προσφύγει στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξετάστηκε στο Ευρωπαϊκό Γενικό Δικαστήριο και τώρα εδώ βρισκόμαστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παρουσίαση μου θα επικεντρωθώ σε δύο τομεί. Πρώτον, θέλω να σα παρουσιάσω ε, την εκστρατεία μας στην Ουγγαρία με την ε, ένωσή μας, την οργάνωσή μας που λέγεται Ράκοτσι και στη συνέχεια θα αναφερθώ στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία μας παρελθούσα και τρέχουσα. Εγώ είμαι νομικό σύμβουλος της ε, Ένωσης Ράκοτσι. Είναι μια οργάνωση κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, ε, ε, που εργάζεται από το 1989 για τι ουγγρικές κοινότητες που ζουν εκτός των συνόρων της Ουγγαρία. και προσπαθεί να συνενώσει αυτές τις κοινότητες με το πληθυσμό εντός της Ουγγαρίας. Έχουμε πάρα πολλά μέλη πάνω από 24.000 και περίπου 500 ε, οργανώσεις τοπικές. Πέρσι το Νοέμβριο όλα τα ουγγρικά πολιτικά κόμματα ε, με κοινοβουλευτική παρουσία υποστήριξαν την πρωτοβουλία αυτή που λέγεται Minority Safe Pack. Επειδή είμαστε ανεξάρτητη ε, οργάνωση μας ανέθεσαν να συντονίσουμε την εκστρατεία αυτή στην Ουγγαρία. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με όσους περισσότερους μπορούμε. Καλέσαμε και τα πολιτικά κόμματα και ε, ε, διαφόρους ενδιαφερμένους, ακόμα και τις εκκλησίες. Για να καταλάβετε, ακόμα και τα ουγγρικά ταχυδρομεία συμμετέχουν από την 1η Φεβρουαρίου. Σε όλα τα ταχυδρομεία υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και μπορεί ο κόσμος να ε, την στείλει ε, στη δική μας ε, οργάνωση. είναι κάτι έντυπα και μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε από πλευρά συλλογή υπογραφών. Έχουμε περίπου 100.000 online και άλλες τόσες ε, χαρτί υπογραφές η λέξη. Στην Ουγγαρία βέβαια αυτή η πρωτοβουλία Minority Safe Pack είναι πολύ ισχυρή στην απήχηση που γνωρίζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ούγγροι που ζουν εκτός της Ουγγαρίας σε γειτονικέ χώρες. Περίπου 2,2 εκατομμύρια Ούγγροι και στην Ουγγαρία έχουμε 13 αυτόχθονες εθνικές μειονότητες που ζουν στη χώρα μας. Αυτό το θέμα είναι πολύ φλέγον και ενδιαφέρει τον κόσμο και προσπαθούμε να τους κινητοποιήσουμε. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Συντονίζουμε τη συλλογή των υπογραφών, κάνουμε εκστρατεία ενημέρωση στον τύπο από τον Δεκέμβριο και μετά. Και τι διαπιστώνουμε. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, δεν γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Και δεν είναι πρόθυμοι. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το πράγμα, περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει στην Ουγγαρία αντίστοιχο εργαλείο, υπήρχε στο παρελθόν. Στην ένωμη τάξη μα δεν έχουμε αυτό το εργαλείο τη πρωτοβουλία πολιτών. Και σου λέει ο πολίτη τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Επίσης, κάτι άλλο ε, που δυσκολεύει τους πολίτες είναι το έντυπο για τη συλλογή υπογραφής. Δεν καταλαβαίνουν. Γιατί σε κάθε έντυπο μπορούν να υπογράψουν μόνο τρεις. Πραγματικά έχουμε μεγάλη δυσκολία δεν το βρίσκουν ε, φιλικό προς το χρήστη αυτό το εργαλείο της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και εγώ το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα. Κάτι άλλο, ε, γιατί ο κόσμος είναι απρόθυμος, δεν θέλουν να δώσουν τον αριθμό ταυτότητας. φοβούνται. θέλει αριθμό ταυτότητας το έντυπο. τι θα ήταν καλύτερο να δώσουν τη διεύθυνσή τους. Αυτό θα ήταν χειρότερο. Θα μπορούσαν να έχουν καταχρήσεις Γενικώ ο κόσμος φοβάται να δίνει τα προσωπικά του στοιχεία. Και για να ε, ασχοληθώ με την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σας πω κάποιες σκέψεις μας. Ορισμένες μας ικανοποιούν ε, από τις προτάσεις. Είναι στο σωστό δρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλην όμως υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που χρειάζονται αλλαγή. Η μερική καταχώρηση είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει ε, και στην περίπτωσή μας ήταν η πρώτη φορά που μία καταχώρηση ήταν μερική και έχουμε και μία κωδικοποίηση. Ε, και μας ικανοποιούν μερικώς επίσης κάποια άλλα στοιχεία της πρώτης. Ας πούμε, η περίοδος συλλογής υπογραφών. Uh, Τρεις μήνες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία. Από την άλλη, η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων μιλάει για 12 μήνες. Κάπου στη μέση θα ήταν ε, ενδεχομένω η σωστή διάρκεια. Όπως βλέπουμε στη δική μας πρωτοβουλία, η συλλογή των υπογραφών άρχισε επίσημα τον Απρίλιο. Αλλά η ουσιαστική εκστρατεία ξεκίνησε αργότερα στην πράξη. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε υπάρχουν λόγοι. Για να μαζέψει υπογραφές χρειάζεσαι ε, πολιτικές δομές. Αυτά τα έχουν τα κόμματα. Η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις της δεν έχουν τέτοιου είδους δομές και δεν είναι προετοιμασμένοι για να συλλέξουν υπογραφές. Οπότε έξι μήνες η προετοιμασία είναι καλύτερη και όχι τρεις. Βεβαίως ε, πολύ καλό είναι αυτό που προτείνουν για την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών, αλλά επίσης συστήνουμε εδώ να ακολουθήσουμε αυτά που προτείνει η έκθεση της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ανεξάρτητο ε, όργανο για τις προτάσεις. Ή άλλες τώρα προτάσεις ε, για τη μόνο απευθυντική θηρίδα και όλα αυτά, one stop shop, εντάξει, να... σκοπός είναι να ενημερώνεται καλύτερα ο κόσμος. Ένα σημείο ακόμα της πρότασης θέλω να αναφέρω και να τονίσω που δεν ξέρω μήπως είναι λάθος το κείμενο. Ελπίζω η πρόθεση να μην είναι αυτή που γράφει εδώ γιατί το δεύτερο σημείο στο άρθρο 12 λέει ότι η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους μόνο εάν συλλέξουν τον απαραίτητο κατώτατο αριθμό υπογραφών. Πολύ κρίμα και λάθος θα ήταν. Δηλαδή, αν σε μια χώρα δεν ε, συλλέξεις τις υπογραφές ε, που προβλέπονται αναχώρα δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ στο ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω, δεν είναι σαφής αυτή η διατύπωση. About the political, the real political impact. Τώρα, ο πολιτικός αντίκτυπος και η συνέχεια που δίνεται. Συμφωνούμε απολύτως με τους προλαλήσαντες και τη δήλωση για την εκστρατεία της ε, πρωτοβουλίας πολιτών. Πρέπει να βελτιωθεί ο πολιτικός αντίκτυπος και το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας υποβάλω μια ιδέα εδώ. Στη σημερινή διατύπωση του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να βγάλει πολιτικά και νομικά συμπεράσματα ε, όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή την νομοθετική πρόταση ή όχι. Τώρα όμως, από τη νομική σκοπιά, αν είναι εντάξει η πρόταση, θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια άλλα στοιχεία και κάποιες άλλες λύσεις. Πώς θα το πω, αν νομικά ευσταθεί κάτι και οι αντιρρήσεις είναι μόνο πολιτικές, τότε μπορεί να είναι προβληματικό αυτό. Αυτό που είπε και ο κύριος Όργαν προηγουμένως. Και θα τονίζω και πάλι την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Για την παραδοχή αυτή που αναφέρει, καλό θα ήταν ε, να ακολουθεί αυτή η και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. And uh, what I already uh, mentioned before και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε γιατί σε κάθε φύλλο ε, μπορεί να υπογράφει ένα συγκεκριμένο αριθμό μέχρι τρεις. Ε, δεν είναι φιλικό προ το χρήστη. Έχουν ένα φύλλο, μια σελίδα και πρέπει να υπογράψουν μέχρι τρει. Μα γιατί μόνο τρει, αφού χωράει παραπάνω. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τάρνοκ. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Ευχαριστώ με τον κύριο Βαλέσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λύνει επαρκώς ε, την αβεβαιότητα που αφορά την ευθύνη των διοργανωτών και ένα πολύ σημαντικό θέμα της προστασίας δεδομένων. Θεωρείτε ότι υπάρχει βελτίωση στον τομέα αυτό. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον υπάρχει επαρκής ενημέρωση ε, μεταξύ των πολιτών για αυτό το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως ε, εργαλείο για συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα εργαλεία εθνικής συμμετοχής. Και τέλος θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας θεωρείται ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των διοργανωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τώρα και εγώ με την ιδιότητά μου ως ε, συντονιστής ε, της ΑΦΚΟ, συγγνώμη, ως εισηγητής της ΑΦΚΟ, όχι ως πρόεδρος. Έχω διπλή ιδιότητα αυτή τη στιγμή. Ε, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπατε στην προηγούμενη διαδικασία. Θα ήθελα να πω ότι η Λετωνική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα ε, χρήσιμη για την έκθεση. Ε, αναφερθήκατε λίγο στη χρηματοδότηση και είπατε ότι ακόμα και αν σας δώσουν 50 cent αρκεί, αλλά τι γίνεται με τη διαφάνεια. Δηλαδή, εάν κάποιος υποβάλει ε, κάτι και σας υποστηρίζει με πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Πόσο ε, διαφάνεια πρέπει να υπάρχει. Δεν χρειάζεται τώρα να σας μιλήσω εδώ για Ρωσία, fake news, ε, αμφίβολα ποσά, προέλευση ποσών μάλλον. Δεύτερον, δεν μας είπατε τίποτα για το πώς ανταποκρίνεται το Λετωνικό Κοινοβούλιο σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Πόσο δημοφιλείς είναι αυτές οι προτάσεις. Μας είπατε ότι το 50% ε, συζητήθηκαν στη Βουλή, αλλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή φτάσουν σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Τρίτη ερώτηση, από περιέργεια. Πώς ε, σας ήρθε η ιδέα Νομίζω ότι το λετονικό εργαλείο είναι το πρώτο, είναι ακόμα πριν και από το φιλανδικό. Πώς σας ήρθε η ιδέα, έτσι από περιέργεια ρωτάω. Και θα ήθελα να επιβεβαιώσω και την εντύπωσή μου ότι η πρακτική της Λετωνίας είναι πολύ πιο ευέλικτη από αυτό που έχουμε εμείς εδώ στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον διότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη εκτός και αν πρέπει να είναι τα πάντα πολύ πιο αυστηρά ελεγχόμενα στην ευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά αυτή ίσως είναι συζήτηση για άλλο θέμα. Τώρα, στον κύριο ε, Γκούντρια, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το δικαίωμα στο νερό ε, που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε πώς θα καταφέρατε, γιατί είναι η μόνη πρωτοβουλία που ήταν ε, επιτυχής σχεδόν. Τίποτα δεν είναι τέλειο βέβαια. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι αυτή. Δεύτερον, το θέμα του ελέγχου των υπογραφών. Υπάρχει το λεγόμενο πρόβλημα Mickey Mouse, ότι μπορεί να έχετε πάρα πολλές υπογραφές ε, ε, με το όνομα Mickey Mouse ή Donald Duck. Κάπω πρέπει να ελέγχετε το υπογραφέ. και αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο πρόβλημα. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να σας πω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά δεν είναι φιλιππόκος ε, παράγων και ε, διευρύνει το, το χώρο στον οποίο ε, ελέγχει τα πράγματα, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι και δικλείδες ασφαλείας και αυτό γίνεται και στις Βρυξέλλες. Τώρα, κύριε Τάρνοκ, ε, να σα πω ότι ναι, προσπάθησα να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει και τη δυνατότητα να απαντήσει, να το συμπεριλάβουν. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουν ήδη και δεν νομίζω ε, ότι κάνω λάθος. Θεωρούν ότι είναι παραβίαση ε, της ε, διαδικασίας της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ποιο θέλει το λόγο, κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς τον καθηγητή Κούντριαν. Επανέρχομαι σε αυτά που είπα προηγουμένως ε, σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει η πρωτοβουλία να καταστεί παιχνίδι παρότι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη στο να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την πρωτοβουλία Right to Water, το δικαίωμα στο νερό. Αυτή ήταν μια καταπληκτική πρωτοβουλία. Ε, στην Ιταλία συμμετείχα και εγώ ε, στον αγώνα ε, δημοψηφίσματος για το νερό. Ένα παρεμφερές δημοψήφισμα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι είχαμε το δικαίωμα ε, στο νερό, ε, δημοψήφισμα στην Ιταλία, δημοψήφισμα στην Ελλάδα, η ιδιωτικοποίηση του ε, νερού πώς θα συνεχιστεί σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές. Όλα αυτά τα δημοψηφίσματα είναι βέβαια κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, ε, το μνημόνιο, η λιτότητα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία επιμένουν συστηματικά στο ότι είναι απαραίτητο να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας ε, των υδάτων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω λιγάκι την δική σας την άποψη δόκτωρα Γκούντριαν γιατί αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τελικά αυτά τα οποία κάνουμε εμείς εδώ είναι απλά κουβεντούλα γιατί κατ' ουσίαν το σημαντικότερο είναι όπως σας είπα αυτές οι πρωτοβουλίες για το νερό που έλαβαν χώρα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε ένα θέμα ευελιξίας. Στην περίπτωση του κυρίου Τσάκη θα πάρει το λόγο τώρα εκπρόσωπός του για τρία λεπτά. Uh, Ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματος ε, της πρωτοβουλίας Minority Safe Pack. Εγώ είμαι Ευρωπαίος συντονιστής αυτής της εκστρατείας και ο κύριος Τάρνοκ ε, μίλησε για τις εμπειρίες στην Ουγγαρία αυτής της εκστρατείας. Εγώ θα ήθελα τώρα να πω ε, δύο λόγια έτσι γενικότερα ε, για την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μάλλον, η δική μας πρωτοβουλία στόχο έχει να υπάρξει νομοθεσία για να προστατεύονται οι αυτόχθονες εθνικές μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στις 3 Απριλίου καταχωρίστηκε η πρωτοβουλία μας και έχουμε ένα μήνα για να συλλέξουμε τις υπογραφές μας. Ε, ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα, ακούγοντας και έχοντας ακούσει όλους τους ομιλητές. Η ευθύνη των διοργανωτών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Υπό ποια έννοια. Οι πολίτες που υπογράφουν τις δικές μας αναφορές ή την πρωτοβουλία μας έχουν ψηλές προσδοκίες γιατί τους τάζουμε κάτι. Τους λέμε κάντε το α ή μην κάνετε το β γιατί περιμένουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προτείνει νομοθεσία. Αυτό τελικά μπορεί να έχει διπλή έκβαση. Από τη μια αν ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θετικά ε, προβεί σε νομοθεσία είναι η καλή περίπτωση και άλλη είναι να πει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε δεν πρόκειται να δώσουμε συνέχεια. Αυτό ε, έχει ένα στοιχείο ευθύνη για τους διοργανωτές. Τι θα βγουν να πούνε στο 1 εκατομμύριο ή στο 2 εκατομμύρια υπογράφοντες, γιατί δεν κατάφεραν να έχουν κανένα αποτέλεσμα παρά την ε, προσπάθεια αυτή. Θα ήθελα να ε, απευθύνω λοιπόν έκκληση ε, στην κοινή ευθύνη που έχει το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στους πολίτες που υπογράφουν μια τέτοια πρωτοβουλία, η αναφορά. Θα πρέπει να ε, περιμένουν οι πολίτες, γιατί περιμένουν να βγει κάτι από όλα αυτά. Καλό είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κοινού και να έχουν την ευκαιρία να έχουν και λόγο σε, στα ευρωπαϊκά ζητήματα και να θέτουν τα θέματα στην ημέρα διάταξη. Αλλά αν δεν ακολουθείται από νομοθεσία, τι να την κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία και την εκστρατεία στην Ευρώπη. Ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό. Ένα συγκεκριμένο τώρα στοιχείο για ε, τις επιγραμμικές υπογραφές και αναφορές. Ο κόσμος, οι πολίτες δεν κατανοούν ότι Έχουμε ταυτόχρονα και online και έντυπες υπογραφές. Στην ιστοσελίδα βλέπουν απογοητευτικούς αριθμούς και από την αρχή δεν απέχουμε πάρα πολύ από το 1 εκατομμύριο και λέει ο κόσμος γιατί να υπογράψω έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Αλλά δεν ξέρει ο κόσμος ότι συνεχίζουμε να μαζεύουμε υπογραφές και σε έντυπα και μπορεί να είναι αρκετά ψηλός ο αριθμός σε σχέση με τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Δεν έχουν καμία ενημέρωση γι' αυτό. Ε, άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνουμε τους πολίτες ότι εκτός από τη συλλογή στο διαδίκτυο συνεχίζεται και με την παραδοσιακή μέθοδο. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές απαιτήσει, είναι γεγονός ότι τρεις υπογραφές να εντυπώ δεν είναι πολλές. Αλλά δεν υπάρχει και νέο σύστημα στοιχείων που πρέπει να δίνουν. το, δεδομένα δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία σε άλλες χώρες ζητάνε περισσότερα, σε άλλες λιγότερα, δεν υπάρχει νέο σύστημα και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για τους διοργανητές. Και χρειάζονται 7 ε, πρόσωπα για να αρχίσει μια πρωτοβουλία. Εφτά από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν ολόκληρη εκστρατεία, χρειάζονται ε, να υποστηρίζονται από ε, ισχυρές οργανώσεις, ΜΚΟ, δηλαδή ενδεχομένως και αυτή η ιδέα να χρειάζεται επανεξέταση. Αρκούν 7 πρόσωπα, μήπως ΜΚΟ δεν μπορούν να αρχίσουν μια πρωτοβουλία ως οργανισμοί. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς? Okay, Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στους ομιλητές για σύντομη απάντηση. Ξέρετε εσείς με τον γρήγορο τρόπο που μιλάτε. Δεν χρειάζεται να εξαντλήσετε τα δύο λεπτά και ένα και θα σας φτάσει. Κύριος Μπρένταξ. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε τα οικονομικά και τη διαφάνεια. Και εδώ θα ήθελα να ε, σταθώ και στην ερώτηση για τη Ρωσία διότι ούτως ή άλλως ε, ε, χαρακτηρίζει την περιοχή. Όσον αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης, ε, σαφώς και αναγνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Και ευτυχώς μπορούμε να επιβιώσουμε ακόμα και αν ξεκινήσει η εκστρατεία όλη η Λετωνία εναντίον μας και το περασμένο τρίμηνο αυξήθηκαν ούτως ή άλλως αυτές οι μάχες εναντίον μας γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Καταρχάς, πολύ μεγάλες δωρεές. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες δωρεές. Το πιο μεγάλο ποσό που μπορεί να λάβουμε είναι χίλια ευρώ, το οποίο δηλώνουμε αμέσω δημοσίως ότι το λάβαμε, για ποιον και για ποιο λόγο. Και για μας το να έχουμε πληροφορίες είναι ζωτική σημασίας. Ε, ταυτόχρονα βεβαίως ε, το κράτος ε, ρυθμίζει τι θα πρέπει να αναφέρει μη κυβερνητική οργάνωση στη Λετωνία και κάθε χρόνο ελεγχόμαστε, δηλώνουμε τι δωρεές λάβαμε, τι τις κάναμε κλπ. Ταυτόχρονα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ή μάλλον να τα πω αλλιώς, να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή αν υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα που θέλει να ε, κάνει μια πρόταση, ζητάμε δωρεά χιλίων ευρώ, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε το πόσο χρησιμοποιούν ε, τα πολιτικά κόμματα ε, την πρωτοβουλία μας. Για τους πολίτες τα πάντα είναι δωρεά και πρέπει να είναι δωρεάν, αλλά για τα πολιτικά κόμματα, κυρίως για το μάρκετινγκ, τους ζητούμε να υποστηρίξουν τις υποδομίες μας και μας έχει βοηθήσει ουσιαστικά, γιατί από τις 300 πρωτοβουλίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, στιγμή ανοιχτέ, μόνο 15 είναι από πολιτικά κόμματα και επιχειρήσει. Επομένω υπάρχει αυτό. Το γεγονό ότι καταφέραμε με επιτυχία να κρατήσουμε χαμηλά ε, το ποσοστό τη δική του συμμετοχή. Όταν ένα κόμμα ή μια επιχείρηση δίνει χίλια ευρώ ως δωρεάν, το, δωρεά, το δηλώνουμε δημοσίως. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, διατηρήσουμε την, αυτή τη δομή της δωρεάς, διότι το κράτος λέει ότι η δωρεά είναι κάτι δεν, για το οποίο δεν μπορούμε να ζητήσουμε πολιτική επιρροή. Δεν πουλάμε χώρο, αν ένα πολιτικό κόμμα μας δώσει τα χρήματα θα τα δημοσιεύσουμε, αλλά δεν το επιθυμούμε. Η διαφάνεια όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό, ο μηχανισμός είναι ότι εμείς δίνουμε το φάκελο με τις υπογραφές και το κείμενο της πρότασης, της πρωτοβουλίας. Το κοινοβούλιο το στέλνει στο Μητρό Κατοίκων για να δει ποιοι είναι εγγεγραμμένοι πολίτες και ποιοι όχι. Ε, συνήθως ε, υπάρχουν μερικές χιλιάδες ε, που δεν είναι σωστές, επομένως έχουμε και ένα αποθεματικό κάποιων εκατοντάδων υπογραφών και μετά από εκεί και πέρα καθορίζεται ε, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να σταλεί αυτό στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Νομικών Θεμάτων, ε, Παιδείας κλπ. Ε, συνήθως ε, το Κοινοβούλιο ψηφίζει για την απόρριψη της πρωτοβουλίας αλλά πολύ σπάνια γίνεται κάτι τέτοιο. Σε γενικές γραμμές το Κοινοβούλιο ξεκινάει τις δουλειές ε, της Επιτροπής τους. Ε, ε, ορισμένες φορές οι Επιτροπές του Κοινοβουλίου καλούν και εμπειρογνώμονε και δεν γνωμοδοτούν μόνες τους. Είναι καλή διαδικασία λοιπόν και μετά υπάρχει η όλη διαδικασία ψηφοφορίας. Η ιδέα ε, ξεκίνησε με το κατά πόσον μπορούμε να ξεκινήσουμε ψηφιακά δημοψηφίσματα. Ε, έγιναν πάρα πολλές δεβουλεύσεις σε ένα εξάμεινο και καταλήξαμε ότι καλύτερα να μην κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα πρέπει να έχουμε σε ψηφιακό επίπεδο ιδέες για νομοθεσία και λειτουργήσε πολύ αποτελεσματικά και σίγουρα είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι από την πρωτοβουλία πολιτών. Το βασικό κανόνας είναι ότι οι προτάσει δεν μπορεί να είναι κατά του συντάγματο κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Μπορεί κάποιο να το ερμηνεύσει είτε πολύ στενά είτε πολύ ευέλικτα. Εμείς βασιζόμαστε συγγνώμη, σε βασικές αξίες ε, και έχουμε πολύ καλή συνεννόηση με το Κοινοβούλιο και είμαστε πιο αυστηροί από ό,τι θα ήταν το Κοινοβούλιο και οι πολίτες εκτιμούν ε, που επιτρέπουμε ε, και τη δημοσίευση πραγμάτων για αλλαγή του ε, συντάγματος. Παραδείγματος χάρη τον αλλάξει ο εθνικός ύμνος δεν θα καταστρέψει τη δημοκρατία οπότε θα δημοσιευθεί. Τώρα για τη Ρωσία. Όντω η Ρωσία χρησιμοποιεί δημοσίω τα μέσα της διπλωματία πολύ καλά. Είχαμε αρκετές ε, ε, δημοσίων σχέσεων εναντίον μας. Συνήθως έχουμε κάτι ε, τέτοιο μια φορά το εξάμεινο. Ορισμένα φορά ε, είναι ασήμαντα και γελία, αλλά ορισμένε φορέ, ιδίω από τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο, μπορεί να είναι και πολύ σοβαρά. Ε, το πιο πρόσφατα ε, ήταν πριν από δύο εβδομάδες, μάλλον το... Ε, yes, thank you uh, for Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ο κύριος Χαουτριάν. Θα αρχίσω back to... Uh, από κάτι που είπατε εσείς, Πρόεδρε για τη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν πάντα έλεγχοι, ε, αντίβαρα. Τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορεί η ασίδωτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Ε, προφανώς θα πρέπει να περιορίσουμε κάπως τις δυνατότητές της. Δεν θα πρέπει να λησποδονούμε ότι ξεκίνησε το Better Regulation, το F για την καλύτερη νομοθεσία, ε, για την αναλογικότητα κτλ. Εμείς έχουμε περιορισμένες δυνατότητες στα χέρια μας, όλοι να τις λάβουμε υπόψη. Ε, ένα από τα ενδιαφέροντα ενδεχόμενα που ανέφεραν και άλλοι είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια πρωτοβουλία να μην μπορεί ενδεχομένω να υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει, να υπάρχει ένα δικαίωμα πρωτοβουλία δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να βασίζεται πάντα στη συμμετοχή των πολιτών. Τώρα δεν θα μπω σε πολύ μεγάλη συζήτηση για τη ιδιωτικοποίηση των υδάτων. Ε, διαφωνώ. Ε, εκτός από την Ελλάδα και ξέρουμε γιατί πρέπει να ιδιωτικοποιήσει εταιρείε υδάτων, γιατί τις το ζητούν και πιέζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι. Στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία ε, ε, και στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, κινητοποίησε τον κόσμο στην αρχή τρομάξαμε πάρα πολύ για τη λογοδοσία, για να δούμε ε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Τελικά ε, δεν το λάβαμε υπόψη. Υπάρχει δυνατότητα ε, να το κάνουμε εμείς. Είμαστε μια μεγάλη οργάνωση συνδικαλιστική. Μπορούμε να το αγνοήσουμε, αλλά ο Ευρωπαίος πολίτης θα φοβάται. Προστασία δεδομένων δεν έχω άποψη γι' αυτό. Δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Και εκτός από τους πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών <clears throat> υπάρχει επίγνωση και γνώση γενικά για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών <clears throat> και συχνά μας απασχολεί όταν έχουμε ένα θέμα να το κάνουμε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ή όχι. Βέβαια παραμένει εμπόδιο για πολλές οργανώσεις συλλογή υπογραφών και οι πόροι ε, που δεν έχουν οι οργανώσει. Βεβαίως, ε, τη συνέχεια που θα δίνεται, αν είναι παιχνίδι, αν είναι συμβολικό, αν έχει κάποια σημασία, το να κάνει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αν δεις ότι μετά από πέντε χρόνια επέτυχε, μετά από δύο χρόνια είχαμε τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα μια πενταετία μετά έχουμε την οδηγία για το πόσιμο ε, νερό Πολλέ οργανώσεις που έχουν μικρότερες δυνατότητες και λιγότερα μέσα θα αναρωτηθούν αν αξίζει τον κόπο τέτοια ταλαιπωρία και τόσο χρονική η καθυστέρηση. Ε, εμείς ε, ε, Έχουμε δική μας πλατφόρμα, δεν έχει αρχίσει τη λειτουργία της η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο και το, πρόγραμμα, το πρόβλημα όπως είπατε ότι πολλοί υπογράφουν ως Mickey Mouse, Donald Duck αυτό νομίζω δεν είναι, είναι περιφερειακό το θέμα. Στη Γερμανία είχαμε πάρα πολλές υπογραφές και εμείς ε, φιλτράραμε τις ε, απαντήσεις, τα ε, γραπτά έντυπα και οι συνάδελφοι και τους βγάλαν έξω αυτούς. Γιατί αν πάει στις αρχές γι' αυτό και το ελέγξουν, θα αφαιρέσουν τον αριθμό των υπογραφών που είναι ε, πλαστά πρόσωπα που υπογράφουν ως, ως Mickey και μετά ε, το ανάγουν και στην υπόλοιπη ε, πρωτοβουλία και αφαιρούν τα ονόματα αναλογικά. Χρηματοδότηση εμείς από τα μέλη μας ε, και από τη Συνομοσπονδία Συνδικάτων δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότηση και συλλογής. Εμείς πάντα διαφανείς είμαστε στη λειτουργία μας ε, στα συνδικάτα ε, μας δίνουν πόρους και οικονομικούς και ε, ανθρώπινους και ενημέρωση διαδίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ιστοσελίδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάναμε σήμερα crowdfunding περισσότερο συμμετοχική χρηματοδότηση για να είμαστε και σε επαφή με τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και υπογράφουν είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπο και να μπορούμε να τους ενημερώνουμε και να λογοδοτούμε. Θα μπορούσε να είχε επιλεγεί από την αρχή αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν ακόμα στάνταρ το crowdfunding όταν άρχισε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Αυτά. Ευχαριστώ. Δεν τελειώσατε. Τελειώσα. Ναι, δεν ήθελα να σας διακόψω. Ο κύριος Τάρνοκ, παρακαλώ. Just very short because θα είμαι σύντομος ε, γιατί συμφωνώ με όσα είπατε και όσον αφορά το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα είναι να εξετάσουμε το όλο πρόβλημα από την προοπτική των πολιτών ε, που βλέπουν ότι ενώ συγκεντρώθηκε ένα εκατομμύριο υπογραφές δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μπορούμε βέβαια να ισχυριστούμε ότι η πρωτοβουλία δικαίωμα στο νερό ήταν ε, η ε, μόνη που είχε ίσως κάποιο αποτέλεσμα. Οι πολίτες αν δούνε ότι δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα ε, τότε θα κάνουν ενδεχομένως ακριβώς το αντίθετο. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά το θέμα αυτό ε, και να κάνει και ένα δεύτερο έλεγχο όταν θα αποφασίσει αν θα καταθέσει την πρόταση ή όχι. Και κάτι άλλο. Ε, όσον αφορά την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών, οι πρωτοβουλίες ε, πρέπει να δούμε από πού έρχονται, από ποια τμήματα μιας χώρας, ε, ποια τμήματα στηρίζουν την πρωτοβουλία. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια ηλεκτρονική εκστρατεία ε, χωρίς να γνωρίζει ότι η εκστρατεία είναι επιτυχημένη, σε ποιο τμήμα της χώρας είναι επιτυχημένη να ξέρει κανείς τι είδους λύσεις μπορούν να προκύψουν. Στην Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, σχετικά με την προστασία των δεδομένων, υπάρχει μια προϋπόθεση καταχώρησης. Όταν ξεκινήσαμε τη συγκέντρωση υπογραφών, έπρεπε πρώτα να, καταγραφεί, να καταχωρηθεί κανείς σε μια εθνική αρχή. Αυτό ήταν ένα επιπρόσθετο βάρος, αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, ίσως να είμαστε και η μόνη χώρα η οποία έχει αυτή την προϋπόθεση της καταχώρησης πριν από τη συγκέντρωση υπογραφών. Και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω και πίσω το λόγο στην Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού και έχοντας ακούσει και την άποψη όλων και των ακαδημαϊκών, πάμε στο δεύτερο πάνελ που έχει σχέση στο τρίτο πάνελ, στο τρίτο πάνελ που είναι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και οι θεσμικές προοπτικές. Ε, και με μεγάλη μου χαρά ε, καλωσορίζω τον κύριο Φων Ρόβερς, ο οποίος θα λάβει το λόγο. Είσαστε από την υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ελπίζω να μπορείτε να περισσείτε 10 λεπτά. Thank Thank Ευχαριστούμε πολύ που μας ε, καλωσορίσατε ε, σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, είμαστε βέβαια στο τελευταίο πάνελ. Ελπίζω παρόλα αυτά να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση. Χαιρόμαστε που είσαστε ακόμα μαζί μας. Ίσως θα είναι η δική μας παρουσίαση. Το ντεσέρ σε ένα πολύ ωραίο γεύμα. Έχουν υπάρξει κάποιες ε, διαμαρτυρίες ε, που αφορούν ε, θεσμούς ε, αλλά και άλλες ε, οργανώσεις με γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από την αντιμετώπιση των προσφυγών, ο διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιεί και το δικαίωμα της ανάλυσης πρωτοβουλίας που σημαίνει ότι η διαμεσολαβητής μπορεί να ξεκινήσει και μόνη της έρευνες. Έχουμε πρωτοβουλίες και διαμαρτυρίες που έχουν σχέση και με το ECI νομίζω εσείς ε, είχατε σχέση έτσι κάπως με τις μειονότητες. Πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, οι ε, προσφυγές αυτές αφορούν διαδικαστικά θέματα, παραδείγματος χάνει θέματα που έχουν σχέση με την ε, περίοδο συγκέντρωσης, το χρονικό διάστημα συγκέντρωσης υπογραφών, αν είναι ένας χρόνος ή παραπάνω. Και έχοντας εξετάσει αρκετές τέτοιες ε, ε, προσφυγές, η διαμεσολαβητής ε, αποφάσισε να ελέγξει την διαδικασία, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή λοιπόν η έρευνα έκλεισε το 2015 με προτάσεις για βελτίωση. Και πριν μπω σε αυτά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές που ισχύουν για, το, τη διαμεσολαβητή. Η πρωτοβουλία ε, προβλέπεται στο τμήμα εκείνο των συνθήκων όπου γίνεται λόγος για δημοκρατικές αρχές. Περιγραφείται ως ένα εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας και το ECI αποτελεί ένα ειδικό τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη δημοκρατία δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως στόχο να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης υπάρχει ένα κομμάτι της συνθήκης για τις δημοκρατικές αρχές, όπου γίνεται λόγος και για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Οι πολίτες συμμετέχουν και εκπροσωπούνται ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την άποψη της διαμεσολαβητού ε, θα ήταν λάθος ε, να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην συμμετοχική δημοκρατία και το ECI. Και τα δύο συμπληρώνουν τη δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του ECI. Η διαμεσολαβητή θεωρεί ότι μέσα από το ECI οι πολίτε θα πρέπει να αισθάνονται ότι όχι μόνο ακούεται, αλλά εισακούεται η άποψή τους και κατόπιν τούτου οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη στη δημοκρατική νομιμότητα των ενωσιακών θεσμών. Φτάνω λοιπόν σε προτάσεις για βελτίωση που κατατέθηκαν πρώτα απ' όλα εκείνες που έχουν στόχο τη διευκόλυνση του, του ECI, ε, μετά θα αναφερθώ στη συμμετοχή. Όσον αφορά τη φάση της προετοιμασίας, η ανησυχία της διαμεσολαβητού ήταν να μην υπάρχει ένα ECI ε, το οποίο ε,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 θα αφορά τον ενωσιακό νόμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές και ε, συμβουλές ε, χωρίς να ε, προσκολάται σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις η διαμεσολαβητής προσέθεσε θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεργατική πλατφόρμα. Αυτό ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου μπορεί να βοηθήσει σε θέματα του παραδεκτού. Εάν απορριφθεί η πρώτη πρόταση για το ECI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει παρόλα αυτά να παραμείνει συνεπής. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι σαφές στους πολίτες γιατί η πρωτοβουλία τους είναι απαράδεκτη και να μην υπάρχει σύγχυση μέσα από το Eurospeak. Η μεσολαβητής, από κοινού με άλλους πρότεινε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τους κινδύνους ε, αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη νομικής προσωπικότητας ε, προκαλεί ανησυχίες. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, ε, εξετάζει όλες αυτές τις διατάξεις και όλα αυτά γίνονται και δωρεάν. Υπό τους προτινόμενους κανόνες ε, μπορεί επίσης να υπάρξει μια νομική υπηρεσία που να εξετάζει διάφορα στοιχεία της διαχείρισης της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβανομένης και και δηλώσεων υποστήριξης. Ε, πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια έρευνα και προτείναμε να υπάρχει περίοδος κέντρωση υπογραφών 12 μηνών, η οποία θα ξεκινάει την ημέρα που επιλέγουν οι οργανωτές και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως σημείο κίνησης στους τρεις μήνες από την ημερομηνία καταγραφής. Όσον αφορά την βελτίωση της ικανότητας των πολιτών να συμμετέχουν εν μέρη στα ECA, η Δήμεσολαβητή έχει μια σειρά προτάσεων. Την πιο σημαντική είναι, πιστεύουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε ECI επιγραμμικά. Η πρόταση αναφέρει ότι όσον αφορά την ε, κεντρική συγκέντρωση υπογραφών, αυτό θα πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την, ε, τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπογράφουν μια πρωτοβουλία ECI σε όποιο άλλο κράτος μέλος το επιθυμούν. Για να υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά πρέπει να είναι απλή συγκέντρωση των δεδομένων και αυτό προτείνει η ίδια Μεσολαβητής. Όσον αφορά τώρα τις ε, επιπτώσεις και εκεί η ίδια Μεσολαβητής ε, ε, έχει να κάνει προτάσεις. Μία πρόταση είναι μια δημόσια ακρόαση που να οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή ως μια δημοκρατική δράση ε, για να καλυφθούν οι υψηλέ προδιαγραφές, ε, η δημόσια συμμετοχή και η διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ε, η διαμεσολαβητή πρέπει να έχει ως στόχο η δημόσια συζήτηση να είναι όσο πιο διαφανής γίνεται. Η διαμεσολαβητή προτείνει εκτό από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμμετέχει σε αυτή την ακρόαση. Ε, το Συμβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα ε, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς τη γενική εικόνα, αυτήν κυρίως να έχει κατά νου. Τέλος, ε, η Μεσολαβητής προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτό το χρονικό περιθώριο των τριών μηνών. Δεν φτάνει για να προετοιμαστεί μία ανακοίνωση. Η Κομισιόν προτείνει η περίοδος αυτή να επεκταθεί από τρεις σε πέντε μήνες. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα της διαδικασίας του ECI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, θεωρήσει ότι μια νομική πράξη δεν είναι μόνο, το μόνο μέτρο ε, σύγκλησης και κρίσης ε, ε, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα από την οποία μπορούν να ξεκινήσουν και περισσότερες συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, αναφέρει περισσότερο τη δική της την άποψη, να αναγνωρίσει την επιτυχία, ο κανονισμός αυτή τη στιγμή γνωρίζει μόνο εκείνες τις πρωτοβουλίες όπου έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αλλά ε, πρέπει να αναφέρονται και άλλα ορόσημα. Ε, στην επίσημη απάντησή τη σε μια ECI που έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφέ, η Κομισιόν θα πρέπει να εξηγεί τι πολιτικέ τη επιλογέ με λεπτομέρειε και με διαφανή τρόπο. Παρότι οι πολιτικέ επιλογέ μερικέ φορέ είναι δύσκολε, τέτοιου είδου επιλογέ, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλου, αλλά οι πολίτε του αξίζει να του λένε την αλήθεια. Και τέλο, για τη διαμεσολαβητή είναι σημαντικό ε, οι πρωτοβουλίες να κρίνονται ως ένα εργαλείο για τους πολίτες, η Κομισιόν να κάνει περισσότερο για τη χρηματοδότηση, ε, για τους χορηγούς ε, και οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει να εξετάζεται. Η διαμεσολαβητής αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει και ελέγχους ποιότητας και να ελέγχει και την συμμόρφωση. Ε, η διαμεσολαβητή θα συνεχίσει να ελέγχει τη διαδικασία και όταν οι νομοθέτες θα έχουν αποφασίσει για τους νέους κανόνες, όλα αυτά θα εξεταστούν με κριτικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και με ιδιαίτερη χαρά τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κίνγκα Γιώ που είναι συντάκτης, ε, γνωμοδότησης, συντάκτρια από την ε, ΕΟΚΕ. Και δεν είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο να έχουμε αυτή τη συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας δίνω μέσα στο λόγο. Thank you so much. Thank you, Chair. Um, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Ε, πραγματικά συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα θέματα, αλλά δεν ε, είναι σύνηθες να έχουμε τη φυσική παρουσία εκπροσώπου του οργάνου μας. Πολύ σημαντική συζήτηση ε, σήμερα και θίγει ουσιαστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ε, διάλογος, ε, συμμετοχή και αυτά είναι και στην καρδιά της δικής μας αποστολής στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, το θεσμικό μου όργανο ήταν ε, ακρεφνής υποστηρικτής ε, της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και ήμασταν οι πρώτοι που εγκρίναμε τη γνωμοδότηση από την αρχή στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 14 Μαρτίου στην Ολομέλειά μας. Ήδη υπάρχει το σχέδιο γνωμοδότησης. Αν θέλετε, διατίθεται και αντίτυπα στην αίθουσα μαζί με τον δόκτωρα Τζέιμς Όργαν, τον εμπειρογνώμονα μου που μίλησε και προηγουμένως, Έχουμε κάνει διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιτροπής των Περιφερειών, της Διαμεσολαβητρίας και βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προετοιμάσουμε και να συντάξουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ακόμα από τον περσινό Δεκέμβριο η μελέτη μας, η ομάδα εργασίας μάλλον, έκανε δημόσια ακρόαση έτσι ώστε να κάνουμε πρόταση ε, όπου να εντοπίζουμε τις ε, ιδιαιτερότητε, τα ισχυρά σημεία και τι αδυναμίες τη νέα πρόταση, για να, γνωρίζουν καλύτερα και συμμετέχουν καλύτερα οι πολίτε. Τώρα είναι σε ένα κρίσιμο πολιτικό σταυροδρόμι η πρωτοβουλία πολιτών. Καλωσορίζουμε την πρόταση που ήρθε τόσο γρήγορα μετά την ανακοίνωση από τον πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φραν Τίμερμαν, στην ετήσια διάσκεψή μας ε, για την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού. Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καλωσορίζουμε τη νέα πρόταση ε, που σε μεγάλο βαθμό απλουστεύει τις τεχνικές δυσκολίες που είχαν συνδεθεί με την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, η ε, ομάδα διοργανωτών μπορεί να επιλέξει πότε θα αρχίσει να συλλέγει υποστήριξη και μπορούν ε, να ε, συστήσουν ένα νομικό πρόσωπο για να περιορίσουν την ποινική τους ευθύνη. Ε, επίσης υπάρχει μια συνεργατική πλατφόρμα επιγραμμική μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζουν οι πολίτες ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη μετάφρασης που παρέχουμε εμείς από την ΟΚΕ σε όλους τους διοργανωτές από το 2015. Ωστόσο προτείνουμε ε, εδώ να συμπεριληφθεί και η μετάφραση των παραρτημάτων. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να συμμετέχουν περισσότερο τα κράτη-μέλη, ο ρόλος των οποίων μέχρι τώρα ήταν αμυγός τεχνικός. Επίσης, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ε, μονίμως ε, την πλατφόρμα για να γίνεται δωρεάν η συλλογή ε, των υπογραφών και δεσμεύεται να ενημερώνει καλύτερα το κοινό. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι δεν ανταποκρίνεται πλήρως ένα από τα βασικά αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών η νέα πρόταση. Το είπαν αυτό πολλοί ομιλητές. Να υπάρχει ισχυρή δηλαδή συνέχεια που να δίνεται και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και μεγαλύτερη προβολή η Επιτροπή μας θέλει να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα θεσμικά όργανα, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους διοργανωτέ, να έρχονται, να συζητούν, να παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίε τους. Εδώ είμαι αποχρεωμένη να τονίσω ε, ένα παράδειγμα επιτυχίας ε, από το δικό μου θεσμικό όργανο. Όπως γνωρίζετε, η ΕΟΚΕ. Ε, προσκαλεί διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών σε διάφορες συζητήσεις που κάνουμε, θεματικές ενότητες, ε, στην ομάδα ECA, ακόμα και στην Ολομέλεια. Είτε για να συζητήσουμε την ίδια την πρωτοβουλία, είτε να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να ακολουθούν αυτό το παράθυμα και να δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες και βήματα διαλόγου κατά τη διάρκεια των εξτρατιών και μετά Δεν τελειώνει η εκστρατεία και η δουλειά με μια επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ακούμε από την κοινωνία των πολιτών θέλουν να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι επιτυχεί πρωτοβουλίε να συζητούνται στην Ολομέλειά σας για να δοθεί και μια πολιτική διάσταση και ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρο. Επίση, συστήνουμε να ε, υπάρχει εγγυημένη ε, μια διαίρεση, μια κατανομή αρμοδιοτήτων και ένας ε, επιμερισμός ε, εξουσιών για να μην έχουμε επικαλύψεις. Σήμερα όλα τα χαρτιά στα χέρια της τα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει και εκφύσεως είναι διαμεσολαβητής ε, αυτών των προσπαθειών. Γι' αυτό Υποστηρίζουμε τόσα όσα ζήτησε η κοινωνία των πολιτών και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός διοργανωτής ε, δημοσίων ακροάσεων με παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αντίστοιχο και κατάλληλο υπηρεσιακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, τεκμηριώνει την κάθε, της, ε, αρνητική απόφαση και απόρριψη, είτε αυτή είναι μερική είτε είναι ολική. Καλωσορίζουμε την πρόταση επίσης να επιτρέπεται μερική καταχώρηση. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει η ενιαία και μοναδική απόφαση να παραμείνει γιατί δεν ε, έχουμε εγγυήσεις για τη διαδικασία αν γίνεται σε δύο φάσεις ή δύο στάδια. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία πολιτών για την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η περίοδος αναθεώρησης θα πρέπει να παραμείνει στην τριετία για τον κανονισμό και να μην γίνει πενταετία όπως λέει η σημερινή πρόταση. Τέλος θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι η ΟΚΕ ε, με περηφάνεια ε, ήταν από την αρχή στο πλευρό αυτής της προσπάθειας και θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, Πολιτών. Χάρη στην ετήσια αφιερωμένη στην πρωτοβουλία ε, διάσκεψη που οργανώνουμε χωρίς διακοπή από το 2012, ακόμα και σε καιρούς που δείχναν οι άλλοι κάποια προθυμία, αυτό δείχνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε σε υψηλή προτεραιότητα αυτό το εργαλείο. Ελπίζουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι ε, θεσμικά όργανα να αναγνωρίζουν τη σημασία της ΟΚΕΔΟ και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, το ECI Day, την ημερίδα αυτή, τις μεταφράσεις, ε, τις δημοσιεύσεις και άλλα εργαλεία online. Εμείς ποντάρουμε σε αυτή την ημερίδα την ετήσια για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για ενημέρωση και για καλύτερη λειτουργία. Επ' θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους στη φετινή μας ημερίδα, η οποία θα λάβει χώρα στις 10 Απριλίου στο κτίριο της ΟΚΕ και ήδη μπορείτε να βρείτε εκτός της αιθούσης ε, τα ενημερωτικά φυλάδια. Προτείνουμε λοιπόν να προσκαλείτε πάντα στις δημόσιες ακροάσεις Επιτροπή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ε, μας ε, συμβουλεύεστε όταν κάνει προτάσεις αναθεώρηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε ε, στην ακροασή σας ε, μετά από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ολομέλειά μας η δημοκρατία και τα παραδοσιακά της εργαλεία αλλάζουν μπροστά στα μάτια μας καθημερινά. Οι πολίτες θέλουν να έχουν λόγο, όχι μόνο ψηφίζοντας κάθε τόσο, αλλά ε, όταν μια κοινή ε, υπόθεση αφορά τις ζωές τους. Είναι νεαρή ε, σε ηλικία αυτή η πρωτοβουλία ως εργαλείο, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει να σταθεί στα πόδια της και να αποτελεί ένα εργαλείο διαλόγου πολιτών και θεσμικών οργάνων. Ας μην χάσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία ε, να χειραφετήσουμε τους πολίτες μέσω αυτού του εργαλείου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ρούντινγκ Μπόρκερ, το οποίο είναι από τους ομιλητές που έχουμε συχνά εδώ στην Επιτροπή μας και περιμένουμε να ακούσουμε και σήμερα τι έχετε να μας πείτε. Είναι τμήματάρχης για το πρόγραμμα εργασίας και τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, ε, ακούστε προσεκτικά τι έχει να μας πει. Ευχαριστώ πολύ για την ε, λαμπερή παρουσίαση και σας ευχαριστώ καταρχάς που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την πολύ χρήσιμη συνεδρίαση και ακρόαση. Ευχαριστώ επίσης και για τη συμβολή τους όλους εκείνους που μίλησαν και νομίζω ότι τις απόψεις τις γνωρίζαμε, αλλά πάντα μπορούμε να δούμε και κάποια πράγματα από διαφορετικό πρίσμα, επομένως σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο να ανατρέξω ε, στα βασικά θέματα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, το βασικό πυρήνα που θέλει να βελτιώσει και ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, έχει δηλώσει δημοσίως ότι θέλουμε η πρωτοβουλία των πολιτών να είναι πιο προσβάσιμη, λιγότερο επαχθής και εύκολη στη χρήση της για τους πολίτες και τους υποστηρικτές και είναι όλοι μα ε, κατά καιρού και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις πλήρε δυνατότητε τη πρωτοβουλία να τα προχωρήσουμε αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Αυτά είναι και τα δύο ε, στοιχεία που μας καθοδηγούν και νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, οι πρωτοβουλίες να καταχωρίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να φτάνουν το κατόφλι του ενός εκατομμυρίου και φυσικά να έχουν και τις μεγαλύτερες δυνατότητες να προχωρήσουν στη συνέχεια. Αυτά είναι τα βασικά. Και να πω το εξής. Πρώτα-πρώτα ε, και θα ήθελα ως υπάλληλο τη Επιτροπής ε, να πω ότι δεν είναι μόνο καθήκον μου αλλά είναι και θέμα προσωπικής ακεραιότητας να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για αυτή την πρωτοβουλία, θέλει να είναι επιτυχής ε, και το έχει αποδείξει όχι μόνο στην πρότασή μας αλλά και από τις πράξεις μας μέχρι τώρα. Κάποια από τα νέα στοιχεία που προτείνουμε είναι ότι ελάχιστοι το σχολίασαν αλλά θέλουμε να μειώσουμε την κατώτατη ηλικία στα 16 που σημαίνει 10 εκατομμύρια ε, πιθανούς ε, ε, επιπλέον πολίτες που θα υπογράψουν. Και το λέω αυτό και με κάποια περηφάνεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολιτικό βήμα και νομίζω ότι όλοι, ελπίζω και τα θεσμικά όργανα και τα συμβουλευτικά όργανα θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και μιλάω εδώ στη γειτόνισά μου εξ αριστερών. Θα λάβετε και ένα σχέδιο κειμένου Δεύτερον, και αυτό είναι στο πρώτο στάδιο και πάλι, θέλουμε να ενισχύσουμε τη βοήθεια προς τους διοργανωτές για μέτρα ε, και βοήθεια στη διοργάνωση. Υπάρχει ε, ένα μητρό για τις πρωτοβουλίες και μια ιστοσελίδα, αλλά θέλουμε να υπάρχει και αυτή η διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα που ε, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει και ως διαμεσολαβητής και ως μέντορα σε κάποιες περιπτώσεις για να βοηθήσει πιθανούς διοργανωτές. Αυτό ε, θα είναι και ένα φόρουμ συζήτησης και να ευχαριστήσω και ε, τον συνάδελφο που συμμετέχει. Ε, προσλάβαμε μια κοινοπραξία που έχει πραγματική εμπειρία και θα μας βοηθήσει πολύ. Θα υπάρχει ένα φόρουμ συζήτησης λοιπόν και θα είναι και ένα βήμα για να ξεκινήσουν κάποιες εκστρατείες με επιτυχία και να δοθούν και νομικοί συμβουλές σε προκαταρκτικό στάδιο και ελπίζω και crowdfunding, δηλαδή ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι βασικό θέμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή πρωτοβουλία και να ξεκινήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης υπάρχουν βελτιώσεις στην ίδια τη διαδικασία της καταχώρησης. Έχουμε προβλέψει ρητά το ενδεχόμενα όταν μια σταλή, μια πρωτοβουλία ε, στην, να μην πηγαίνει στο επίσημο, ε, πιο υψηλό επίπεδο της Επιτροπής, αλλά σε τεχνικό επίπεδο να μας για να μας πούν αν υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε πρώτο στάδιο για να μπορέσουν να τροποποιήσουν, να το σκεφτούν. Ε, δεν θα τους γράψουμε εμείς τι θα πούνε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν μια αναδιατύπωση βάσει των σχολείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα αυξήσει τις, αυξήσει τις πιθανότητες καταχώρησης. Και επίσης υπάρχει και η δυνατότητα μερικής καταχώρησης. Και εκεί έχουμε ήδη κάνει αυτό το οποίο ε, πρεσβεύαμε. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 17 καταχωρήσει και μόνο μία την απορρίψαμε. Ε, υπήρχε κάτι για τον Brexit που ακόμα και ο πιο λαμπρός ε, νομικός δεν μπορούσε να δει τις εξουσίες μας και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μπορούν να ασχοληθούν με το θέμα του Brexit. Επομένως θεωρούμε ότι είναι σχεδόν 100% η επιτυχία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει εφαρμόσει, θέλουμε να το εφαρμόσουμε όμως και στο νέο κανονισμό. Ε, προτείναμε και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το σχολιάσατε ήδη, να υπάρχει μια περίοδος ε, τριών μηνών εντός της οποίας να μπορούν να αποφασίσουν οι διοργανωτές και να δουν τι θα προχωρήσουν. Είναι σημαντικό το διάστημα αυτό διότι υπάρχει και ένα κεντρικό σύστημα ε, συλλογής υπογραφών, ε, το οποίο θα το διαχειρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λαμβάνει υπόψη της και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα είναι υπεύθυνη η Επιτροπή και θα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία αν κάποιο θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Ε, είδαμε και τις συζητήσεις για τα απαιτήσει για τα δεδομένα, τα έχουμε συζητήσει ήδη, τα έχουμε και στο έγγραφο εργασίας το οποίο συνοδεύει την πρόταση και λέμε γιατί μειώσαμε από τα 13 μοντέλα στα 2 μοντέλα μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και εξηγούμε και γιατί είναι το πιο καλό μοντέλο αυτό. Ε, και Φυσικά και τα κράτη-μέλη καμιά φορά πρέπει να κάνουν επαλήθευση αυτών των στοιχείων δεδομένων. Βλέπουμε τι δεδομένα υπάρχουν σε κάποιε χώρε. Υπάρχουν δύο μορφέ. Αυτή είναι η μέγιστη δυνατή απλούστευση που μπορούμε να προτείνουμε, αλλά το κάναμε. Στη διαδικασία τη εξέταση, που είναι αυτό το οποίο συζητήθηκε περισσότερο. Εδώ δεν νομίζω ότι ε, θα κρυφτούμε από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο νομικό και θεσμικό ε, πλαίσιο και πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε και να μην είναι παράνομα αυτά που γίνονται και νομίζω ότι αυτό το αντανακλά η πρότασή μας ε, και θα είναι χρήσιμο, το συζητήσαμε και ελπίζουμε να το συζητήσετε κι εσείς. Λαμβάνω υπόψη μου ότι και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου ήδη έχει γνωμοδοτήσει για το κατά πόσον κάποια στοιχεία θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θεωρεί ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να επεκταθούν. Επομένω, συμφωνεί με την ε, νομική άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζουμε ότι και οι άλλε υπηρεσίε θα έχουν την ίδια άποψη. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε όχι μόνο σε εκείνου που μίλησαν, αλλά και να πούμε στου πολίτε ότι υπάρχει ένα όριο θεσμικά και νομικά, το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό απολύτω, διότι ε, ζούμε εντό του δικαίου. Ε, η όλη μα λειτουργία εξαρτάται από το κατά πόσον σεβόμαστε τον νόμο. Και η Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνθήκων θα είναι η πρώτη που θα το υπενθυμίσει αυτό και δεν θα υπερβεί το όριο προφανώ. Πέραν αυτού όμω, αυτό επί του οποίου συμφωνούμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι υπάρχει εκπροσώπηση και να υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία γιατί υπάρχει δυνατότητα συζήτηση όταν υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ιδάλω δεν είναι πραγματική συζήτηση αυτό που γίνεται. Δεύτερον, έχουμε και το έχουμε προβλέψει και στην πρόταση και παραμένει ε, να κοινοποίησαμε σε όλα τα θεσμικά όργανα και συμβουλευτικά όργανα και την ΕΟΚΕ, τη συνάδελφό μου εδώ στα αριστερά μου, σε κάθε επίπεδο και σε επίπεδο ε, επιτυχίας. Δηλαδή η συμμετοχή μπορεί να είναι εξασφαλισμένη. Και επίσης έχουμε επεκτείνει την περίοδο εξέταση από τους 3 στους 5 μήνες. Υπάρχει περισσότερος χρόνος συζήτησης, αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος της Μεσολαβήτριας εδώ, και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άκουσα πολύ προσεκτικά και υπάρχουν και κάποια θέματα για δυνατότητα επέκτασης του ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτό το στάδιο της εξέτασης, ε, λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα ε, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα παραδείγματα δηλαδή. Και αυτά φυσικά είναι εντό τη εντολή του Κοινοβουλίου, μπορεί το Κοινοβουλίο μπορεί να το συμπεριλάβει αυτό σε κάθε στάδιο, σε πολιτικό επίπεδο βέβαια ε, πρέπει να αναφερθούν αυτά. Καλό ε, θα ήταν λοιπόν και εμείς να τα υποστηρίξουμε. Δώστε μου και δύο λεπτά να αναφέρω σε κάποια σημεία στα οποία ε, αναφέρθηκα ήδη τους περιορισμούς και οι νομικές αλλαγές και νομικές μιας νομικής πράξης. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον ορισμό της νομικής πράξης του Legal Act. Θεωρούμε ότι είναι ο πιο ευρύς ορισμός που έχουμε. Ε, σε κάθε ε, ένομη τάξη θα υπάρχει διαφορετική ε, δυνατότητα. Τα δύο που χάσαμε είναι τα δύο τρίτα. Τα τέσσερα ήταν τα επιτυχή και μας επέτρεψαν να ασκήσουμε τις βασικές μας εξουσίες. Αυτό δεν τα αναφέρει, αλλά είναι τα δύο τρίτα. Πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς λοιπόν για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Και σε αυτές τις δύο υποθέσεις αμέσως ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκανε μερική καταχώρηση της πρότασης. Ε, δεν λέω ότι προφανώς τα πάντα θα πάνε καλύτερα, αλλά ο κόσμος δεν είναι τόσο ζωφερό αν τα δύο τρίτα πηγαίνουν καλά. Μπορώ να σας πω ότι σε κάποια δικαστήρια μπορεί να θεωρηθεί και καταπληκτική επιτυχία. Τώρα, το παραδεκτό. Το έχω ξαναπεί και εδώ, και ως υπάλληλο αλλά και ως άτομο, προσβάλλομαι όταν γίνεται συζήτηση από, ε, για δικαστές και ε, ε ενόρκους το, ο έλεγχος του παραδεκτού δεν ήταν στο σχέδιο κειμένου του αρχικού κανονισμού για την πρωτοβουλία των πολιτών. Συμπεριλήφθη η βάση της συζήτησης και γιατί, γιατί θα ήταν άδικο να ζητήσουμε πρώτα από τους διοργανωτές να φέρουν με ένα εκατομμύριο υπογραφές και μετά τους λέμε «Α, δεν είναι παραδεκτό». Βάλαμε λοιπόν εκ των προτέρων το παραδεκτό και γιατί δόθηκε αυτό το πλεονέκτημα στην Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σαφήνεια και συνέχεια και να συνεχιστεί στη συνέχεια από εκεί και πέρα. Και αν οποιοδήποτε φορέα, οποιοδήποτε είναι, και από ό,τι άκουσα ο διαμεσολαβητή δεν είπε αν είναι ο πλέον αρμόδιο για να κάνει μια ε, ποιοτική αξιολόγηση και όχι μια νομική διοικητική ε, αξιολόγηση. Και νομίζω ξέρω την απάντηση, γι' αυτό δεν κάνω και την ερώτηση. Το θέμα είναι ότι αν γίνεται από κάποιον άλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλο, μετά τη συλλογή του ενό εκατομμυρίου υπογραφών, θα πρέπει να κάνει την αξιολόγησή τη βάσει συνθήκων. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Επομένω, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όσον αφορά το παραδεκτό έχει τον τελικό λόγο για το κατά πόσο θα γίνει παραδεκτό ή όχι ένα αίτημα. Ε, Ίσως λοιπόν δεν θα έπρεπε να σκεφτόμαστε εναλλακτικέ λύσεις γιατί ούτως ή άλλως αυτό προβλέπεται. Τέλος. Η υποχρέωση δράσης όταν γίνει υποβολή μιας πρότασης. Σίγουρα υπάρχει θεσμικό θέμα αυτό. Το συζήτησαν και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν την ε, ε, αρμοδιότητα να το πούνε και αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σε τελική ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει τι διαδικασίε τη πριν προτείνει οποιαδήποτε νομική πράξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το λάβω σοβαρό υπόψη, γιατί είναι τμήμα τη εντολή μου και είναι τμήμα και αρμοδιότητα τη γενική μου διεύθυνση, αλλά θα βελτιώσει σίγουρα τον, νόμο, τον τρόπο που νομοθετούμε. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επικουρικότητα. Και κάποια από τα θέματα που συζητώνται εδώ κάποιες από τις ε, παρατηρήσεις για επιτυχείς πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να ε, ε, γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι υποχρέωσή μας να αξιολογήσουμε για την επικουρικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτομάτως να δεχτούμε ότι αν υπάρχει μια πρόταση πρέπει αυτόματα να μεταφραστεί σε νόμο, γιατί υπάρχουν και όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσει που έχουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνω με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί προ όλου εκείνου που μιλούν με του πολίτε και ξέρω ότι εσεί συνομιλείτε με του πολίτε και να είμαστε ε, έτοιμοι. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μια πρωτοβουλία. Δεν υπήρχε δυνατότητα να είναι κάποιο αντίθετο σε μια πρωτοβουλία. Εάν μεταφραστεί αυτόματα σε νόμο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει τι προβλήματα θα υπάρχουν ε, ως αντίδραση. Αν θέλετε ασφάλεια δικαίου και ισχυρίζεστε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση ε, στη γλυφοσάτ για παράδειγμα, ε, που είναι αυτό το οποίο ζητούσαν οι πολίτες, θα ξεκινήσει αμέσως μια αντίθετη πρωτοβουλία. Και αυτό θα είναι ακόμα πιο προβληματικό για το μέσο, γιατί θα υπάρχει ναι πρέπει να την απαγορεύσετε και όχι πρέπει να την παρατείνετε για 10 χρόνια. Και το θέμα είναι ε, ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε οποιοδήποτε πολίτη θέλει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό θα θέσει εν κινδύνο ε, την όλη διαδικασία. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ε, μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Έχουμε το παράδειγμα της Φινλανδίας για το θέμα των ε, γάμων, ε, του γάμου μεταξύ ε, ομοφιλοφίλων. Και ο κύριος Σόπφλιν τώρα παρακαλώ για να κάνει παρέμβαση ή να θέσει ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις σας για αυτά που μας είπατε. βεβαίως Πάντα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον ε, τα θέματα που μας θίγεται, ε, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ε, μερικές φορές υπάρχει μια εχθρική ατμόσφαιρα, αλλά θα λέγει κανείς ότι αυτό ανήκει και στη δουλειά που κάνετε. Δεν θα αναφερθώ σε όλα που ακούσαμε σήμερα, αλλά θα ήθελα να δείξω ορισμένα θέματα. θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη ε, πρέπει όχι μόνο να φαίνεται αλλά και να υπάρχει. Ε, γίνεται λόγος για ανεξάρτητο φορέα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να παρατηρήσω. Το δεύτερο, ε, η παραδοχή. Το μαχητό τεκμήριο. Κατά κάποιον τρόπο Δεν υπάρχει νομική παραδοχή, νομικό τεκμήριο, παραδοχή μάλλον. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ε, πέσουν όλοι υπογραφές, δηλαδή Μία υπογραφή κοστίζει 1 ευρώ, ίσως με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό που σημαίνει είναι ότι μιλάμε για μεγάλα ποσά τα οποία είναι απαραίτητα και πρέπει να ξέρουμε τις πηγές από που προέρχονται. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ε, και αν θέλετε ε, να ε, μιλάμε για ένα επιτυχημένο εργαλείο και δημοκρατικό εργαλείο. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, το είπα και στον κύριο Τίμερμαν, δηλαδή όταν ερμηνεύετε πράγματα παρακαλώ να έχετε μια γενναιόδορη ερμηνεία, γιατί στο νόμο πάντα υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, μπορεί κανείς να είναι στην ερμηνεία του πιο περιοριστικός ή πιο γενναιόδορος. Κατά το παρελθόν είχα την αίσθηση ότι η Κομισιόν δεν ήταν τόσο γενναιόδορη όσο έπρεπε. Εδώ έχουμε μία ανοιχτή ακρόαση. Πρέπει να σας πω ότι ε, χαρήκαμε που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ε, δεν ξέρω, θα μείνετε εδώ. Ε, αν μείνετε εδώ, καλό βράδυ ή μήπως επιστρέψετε στην Ιταλία. Ο κύριος Γιάρεκ. Κοιτάξτε και εγώ ε, θα πω περίπου το ίδιο όπως και προηγουμένως. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν θα καπελωθεί από ειδικά συμφέροντα ή ας πούμε από τη Ρωσία, Ρωσία φιλική χώρα σε εισαγωγικά. Χρειάζεται να έχουμε τους οικονομικούς πόρους ε, Ε, να έχουμε το νου μας ε, σε οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με το ΙΣΙΑ. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι η εκστρατεία συνειδητοποίησης της κοινή γνώμης ε, Εντάξει, γίνονται εδώ συζητήσει και στην Ολομέλεια, αλλά αυτά αρκούν, άραγε αρκούν ως μηχανισμός για να υπάρχει ε, συνειδητοποίηση. Ξέρω ότι στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συζητάτε και ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά ίσως θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν πιο κατανοητά ε, και να προβληθούν περισσότερο στον απλό άνθρωπο, έτσι ώστε οι μηχανισμοί να είναι πιο αποτελεσματικοί. Ε, δεν ξέρω μπορούμε άραγε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ε, ίσως εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε από αυτό. Νομίζω ότι είναι καλό που γίνονται διάφορες προτάσεις. Ε, θέλετε να τοποθετηθείτε, να πείτε κάτι άλλο πριν επανέλθουμε στους μιλητές. Κυρία Μίτσι, παρακαλώ. Θα ήθελα να θίξω λιγάκι ένα θέμα που αφορά ε, στον εκπρόσωπο από την διαμεσολαβήτρια. Η Κομισιόν έχει κάνει αναφορά στο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αρκετοί άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν πει ότι η διαμεσολαβητής είναι ε, ο σωστός φορέας. Ε, να είναι αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός, ο ανεξάρτητος φορέας που θα κάνει την αξιολόγηση. Δεν ξέρω τι πιστεύει η διαμεσολαβητής γι' αυτό και ε, ίσως μπορείτε να μας πείτε με ναι ή όχι αν Μπορείτε να μας πείτε αν βλέπετε να υπάρχει άμεση συμμετοχή στη διαδικασία για το ECI. Και επίσης ε, η διαμεσολαβητής έχει προσφέρει ε, πάρα πολλές ε, προτάσεις και συστάσεις. Η Κομισιόν έχει πει κάτι που εσείς να πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτές τις συστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας επανέλθουμε λοιπόν τώρα στο πάνελ. Πολύ σύντομα όσον αφορά ε, στο θέμα του να απάγει κανείς ε, την πρωτοβουλία του, να την καπελώσει όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό είναι ένα ερώτημα που προκύπτει συνεχώς ε, στην Επιτροπή μας. Οποτεδήποτε μιλάμε στα μέλη μας που δεν συμμετέχουν σε αυτό το θέμα, το θίγουμε και το συζητάμε. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι εμείς ε, αποτελούμεθα από τους εργοδότες, από τους, ε, τους συνδικαλιστές και από την κοινωνία των πολιτών. Οι άνθρωποι αυτοί γιατί οι εργοδότες είναι εκείνοι που μου είπαν ότι όταν θέλουν να σκίσουν επιρροή ως επιχειρηματίες σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής είναι πολύ πιο εύκολο για εκείνους να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο ε, να προσπαθήσουν να οργανώσουν μια ευρωπαϊκή από το να οργανώσουν μια ευρωπαϊκή κοινωνία, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που είναι πολύ πιο δαπανηρή. Έτσι το βλέπουν το θέμα οι εργοδότες. Τώρα, για τη συνειδητοποίηση αυτό το κάνουμε εμείς. Ε, αυτή τη στιγμή το κάνουμε, απευθυνόμαστε όχι μόνο στους οργανωτές που ήδη συμμετέχουν στην ε, διαδικασία ε, της συγκέντρωσης υπογραφών, αλλά απευθυνόμαστε και στους απλούς πολίτες ε, μπορούν να βρουν πληροφορίες σε, στη γλώσσα τους για το πώς μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν υπογραφές. Είμαστε ανοιχτοί από αυτού του θέματος. Πολύ ευχαρίστως να συνεργαστούμε. Λοιπόν, ε, επειδή εσεί σκέφτεστε τα απαντήσετε, σα πειράζω τώρα να πω εγώ. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος ε, Σόπφλιν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ε, το θέμα δεν είναι μόνο να κάνει κανείς κάτι ή να φαίνεται ότι κάνει κάτι, είναι και να το κάνει στην πραγματικότητα. Όσον αφορά το θέμα του παραδεκτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει ήδη αναφερθεί αυτό, υπάρχει δυνατότητα να καταφύγει κανεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί οποτεδήποτε εκχωρείται μία αρμοδιότητα σε έναν άλλο θεσμό ε, μπορεί κανείς να χάσει αυτό το πολύ σημαντικό δικαίωμα ε, σχετικά με την ε, καταχώρηση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία σταθμισμένη απάντηση κατά την τελική φάση του σχεδιασμού της νομοθεσίας μαχητό τεκμήριο. Νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επ' αυτού γιατί είναι επικίνδυνη ατραπός ε, και ίσως ε, προκύψουν και ορισμένα πράγματα που δεν τα θέλει καν το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη θεσμική ισορροπία. Όσον αφορά τους πόρου. Ε, προφανώς ε, και θέλουμε να υπάρξουν περισσότερες τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Δεν θέλουμε δηλαδή να πρέπει τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τις μεμονωμένες δηλώσεις περί χρηματοδότησης. Επειδή δεν έχουμε στοιχεία, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται καν θέμα η απάντηση της Επιτροπής σε σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι αυτά που υπάρχουν λειτουργούν καλά και δεν έχουμε ενδείξεις για κάτι το αντίθετο. Αν υπήρχε, ε, υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις θα προσπαθούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και μετά τις ανησυχίες μας θα προσπαθούμε να τις μεταβιβάσουμε στην αρμόζια Εθνική Αρχή. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη προσέγγιση αλλά δεν ε, ε, έχει νομική κατοχήρωση γιατί ήδη τις έχουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Και στο σχέδιο ε, προβλέπεται ήδη υποχρέωση των οργανωτών προς ενημέρωση. Εμείς ε, θεωρήσαμε ότι αυτό φτάνει από το να ε, από το να φορτώνουμε το βάρος της οργάνωσης αυτής της πρωτοβουλίας. Να πω και κάτι άλλο. Το 16 και το 17 υπήρχε καταχώρηση, ε, υπάρχει όμως και πολιτική βούληση που καταδεικνύει ότι είμαστε γενναιόδοροι ε, στην ερμηνεία των νόμων. Το Κοινοβούλιο με προτάσεις που έχουν κατατηθεί ε, για να ενισχυθεί η παρακολούθηση ίσως μπορεί να καλέσει την Κομισιόν να λογοδοτήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ε, δεν θέλω να κάνω βέβαια διάφορες κασίες από αυτό γιατί βλέπω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την εκστρατεία συνειδητοποίησης. Ε, ήδη για φέτος ε, έχουμε ενισχύσει αυτή την εκστρατεία για το ECI. Συνεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από την Επιτροπή των Περιφερειών και από εσάς με τα δικά σας τα γραφεία. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εκστρατεία για φέτος, για του χρόνου και ίσως και για το 2020. Κάθε χρόνο χρόνο απευθυνόμεθα σε μια συγκεκριμένη ομάδα κρατών μελών. Έχουμε μια γενική εκστρατεία και μετά είμαστε πιο επιλεκτικοί. Ας πούμε πλησιάζουμε την χώρα που έχει την Προεδρία και τελικά θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ε, απευθυνθούμε και στα 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κυρία Μίτση, και ε, προηγουμένως τα ανέφερε η κυρία Σπινέλη. Αν θα μπορούσε να παίξει ο διαμεσολαβητής ένα τυπικό και επίσημο ρόλο στη διαδικασία. Αυτό έχει συζητηθεί στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού και εμείς είμαστε πολύ επιφυλεκτικοί. Είναι γεγονός ότι αποτελούμε ανεξάρτητο και μη πολιτικό όργανο. ίδια ε, μεσολαβήτρια ε, μπορεί να κάνει πολιτικές δηλώσεις γιατί βρισκόμαστε σε πολιτικό χώρο, αλλά είμαστε ανεξάρτητοι το μη πολιτικό όργανο και έχουμε σαφέστατη εντολή να αντιμετωπίζουμε και να επεξεργαζόμαστε καταγγελίες όταν φτάνουν στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να μας δώσουν ένα ρόλο, να, εξετούμε το, να εξετάζουμε το παραδεκτό μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών και αν ε, στη συνέχεια αυτή οδηγήσει σε καταγγελία μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική. Δεν θα το προτείναμε αυτό να γίνει. Να αναλάβουμε και αυτό το ρόλο. Για την ε, οικονομική διαφάνεια των ε, ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, το είπαμε ξεκάθαρα πέρσι στη δημόσια διαβούλευση και το αντίστοιχο έγγραφο το αρχικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ίδια κατεύθυνση πηγαίνει όπως αυτή που ανέφερε ο δεν έχουμε δει πρόβλημα προς το παρόν με χρηματοδότηση πρωτοβουλειών και δεν έχουμε και κανένα φόβο ή καμία ανησυχία μήπως συμβεί τίποτα στο μέλλον. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Μητρό Διαφάνειας για πώς το αντιμετωπίζει. Υπάρχουν ε, ποιοτικοί έλεγχοι, ε, επιτόπιοι και ένα σύστημα ε, κρούσεις του κόδωνα του κινδύνου και προειδοποίησης. Αν κάποιος έχει υπόνοιες για το παραμικρό, απευθύνεται στη γραμματεία. Και αυτό έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να μην έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πάντως υπάρχει αυτό το σύστημα προειδοποίησης και τα καμπανάκια, εν πάση περιπτώσει. είναι δημόσιες οι δηλώσεις ε, και τα ποθενέσχες και όλα αυτά των ε, διοργανωτών και είναι και πολλά τα μάτια που τα παρακολουθούν και είναι πρόθυμοι να ε, καταγγείλουν οτιδήποτε παράτυπο ή περίεργο συμβαίνει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Now these three interesting hours. Τρεις ενδιαφέρουσες και πλήρεις ώρες ανταλλαγής και συνομιλιών τελειώνουν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για την αντοχή σας. Τρεις ώρες. Όλο το απόγευμα, ακόμα και εσείς το τελευταίο πάνελ, ε, έχετε έρθει από νωρί. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένα θέμα που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την προσοχή πολλών μελών, εμπειρογνωμόνων, ε, ενεχομένων, ενδιαφερμένων και πολιτών που μας ακούνε. Και εμείς είμαστε πάντα εδώ για να τους υπηρετούμε και ποτέ για να τους ε, διατάσσουμε, να τους καταδυναστεύουμε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και να παραθέσω κάποιον ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση πάντα υπάρχει δρόμος και τρόπος να τα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας απόγευμα. Οι συνάδελφοι, εσείς θα πρέπει να παραμείνετε, δεν τελειώσαμε ακόμα.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 are you ready to go? Λοιπόν, έτοιμοι. Πώς τα είπε ο Ομπάμα, έτοιμο, ε, έτοιμος. Yes, I can, απαντάει ο κύριος Βαλέσα. Λοιπόν, για αυτή τη γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ε, είσαι ε, και ξέρουμε τη διαδικασία εάν υπάρχουν κάποια βασικά θυμία τα οποία θα ήθελες να αναφέρεις, να το κάνεις. Αλλά νομίζω ότι περισσότεροι ξέρουμε προς τα που θέλεις να κατευθυνθείς ήδη. Παρακαλώ όμω έχεις το λόγο. Νομίζω ότι τα είπα ήδη προηγουμένως ε, και νομίζω ότι ε, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Να σας πω όμως εν συντομία τι έχω κατά νου σε αυτή τη γνωμοδότηση. Όπως θα θυμάστε, όταν ε, ε ορίστηκα εισηγητής, αρκετές ομάδες εξέφρασαν ε, την επιθυμία να υπάρχει πιο στενή συνεργασία για το θέμα αυτό, κάτι το οποίο αποδέχθηκα ευθύ εξ αρχής ε, ε, και αναζητώντας ε, τη συμβολή όλων των πολιτικών ομάδων ευθύ εξ αρχής, ήδη κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό τον Ιανουάριο, ε, το οποίο δεν γίνεται συνήθως στις γνωμοδοτήσεις. Αυτό όμως αποδεικνύει ότι όντως θέλουμε να έχουμε συμμετοχή ευθύ εξ αρχής για το θέμα αυτό. Περιμένω λοιπόν και στοιχεία από όλους τους συναδέλφους για το θέμα αυτό και εν ώψη και του γεγονότος ότι 1η Μαρτίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η αναθεώρηση της, ε, του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλία των Πολιτών εκρεμεί εδώ και κάποια χρόνια πλέον λόγω ε, κάποιων των ε, δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι πολίτε που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον κείμενο κανονισμό. Και πράγματι αποτελεί και πολύ καλή στιγμή για τη δική μας την Επιτροπή για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Στις 31 Ιανουαρίου έγινε μια τεχνική συνοδρίαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Θεμάτων και της Επιτροπής μας, με στόχο να διευκρινίσουμε περαιτέρω τις πρακτικές και τεχνικές λεπτομέρειες της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ε, συνέχεια είναι, αναμένεται και θα δοθεί το κείμενο στους ε, σκιώδεις μόλις το έχουμε στη διάθεσή μας. Θεωρώ ότι αυτός ο κανονισμός είναι ένας καλός τρόπος να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και το δικό μας το ρόλο, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη συμμετοχική δημοκρατία. Και πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να το κάνουμε. Ε, Κατά την προετοιμασία του πρώτου σχεδίου της γνωμοδότησης ε, έκανα μια προσπάθεια να βρω κοινό έδαφος ε, από προηγούμενες αναφορές και γνωμοδοτήσεις ε, και τις θέσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τη δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας ε, και πρέπει βεβαίως να είμαστε βέβαιοι ότι ε, θα βρισκόμαστε και στην πρώτη γραμμή στο θέμα αυτό ε, την καθοδήγηση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για να είναι η πρωτοβουλία μια, χωρίς αποκλεισμούς και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε. Προφανώς όσο ε, περισσότερο συμπεριλαμβάνει, τόσο περισσότερο σημαντική θα φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία. Αν και πρέπει να το πω. Αν δούμε τη σημερινή ακρόαση και αν εξαιρέσετε και, τη, και εσάς κυρία Πρόεδρε και τους εισηγητές, ήταν ελάχιστοι οι ε, συνάδελφοι εδώ και πραγματικά με στεναχωρεί, διότι ήταν τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση, τόσο ενημερωτική σήμερα και έχουμε μόνο 7 μέλη ε, στην καλύτερη στιγμή μας. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό και θα το συζητήσω και στις συνεδρίες των συντονιστών. Ε, αυτό όμως είναι ε, συνηθισμένο. Κάθε φορά που έρχομαι σε αυτές τις ακροάσεις και οι περισσότερες από αυτές είναι ενδιαφέρουσες, ε, δεν έχουμε αρκετούς ε, συμμετέχοντες και φαίνεται σαν να είναι άχρηστες πια. Ε, να ξανάρθω τώρα στο προκείμενο. Κατά την προετοιμασία της γνωμοδότησης επικεντρώθηκα σε άλλα στοιχεία της πρότασης, το άρθρο 4 για τις ε, ε, πληροφορίες και τη βοήθεια που παρέχεται στους διοργανωτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και το άρθρο 7 που αφορά τη διαδικασία της καταχώρησης. Όπως ε, θα έχετε διαπιστώσει, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πλήρη σε αρκετά σημεία και κάλυψε και κάποιες προτάσεις που έγιναν νωρίτερα στη γνωμοδότησή μας για το θέμα αυτό. Κατά συνέπεια, επέλεξα να επικεντρωθώ κυρίως στους τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικές βελτιώσεις. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όντως περιλαμβάνει τα πάντα και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά μπορούμε και να συμβάλλουμε για να βελτιώσουμε αυτό το σημαντικό εργαλείο. Εξάλλου, όταν θα λάβω όλες τις τροπολογίες ε, θα γίνει και μια συνάντηση με τους κοιόδης συγητές το Μάρτιο. Να σας δώσω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα θα γίνει συζήτηση. προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών 1η Μαρτίου, 3 ε, το απόγευμα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 24 ε, Απριλίου αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα προλάβουμε όλα. Ευθύς εξ αρχής φάνεται ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μηχανισμός και όταν θα έχουμε όλες τις τροπολογίες σίγουρα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλεια Γιάρεκ. Η Μαλένα Μίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλά να πω. Όπως είπε πολύ ωραία ο Γιάρεκ, βεβαίως ε, θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, πρέπει να γίνει εδώ και καιρό και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που πρέπει να βελτιωθούν για την ομάδα των διοργανωτών, για την ευθύνη τους και πώς θα δημιουργήσουν και ένα νομικό πρόσωπο. Και με την επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα και τα σημεία επαφών για τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ε, θα φροντίζει και τις μεταφράσεις. Πολλά είναι τα θέματα ε, στα οποία σε υποστηρίζω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όμως να συγχαρώ τον κύριο Βαλένσα για την εργασία του αυτή, διότι έχετε δημιουργήσει μια εξαιρετική βάση για συζήτηση Και πιστεύω ότι οι τροπολογίε μας και οι δικέ μας και οι δικές σας θα εμπλουτίσουν αυτή την πάρα πολύ καλή βάση ε, συζήτηση που είναι πολύ σημαντική για την συμμετοχική δημοκρατία. Ωστόσο, θέλω λίγο να με ενημερώσετε, παράδειγμα, αυτό που ζητάτε ε, για την offline υποστήριξη και σημεία φυσικής ε, παροχής υπηρεσιών και ε, ε, πληροφοριών και ε, κάποιες υπηρεσίες παροχής συμβουλών προς πολίτες. Δεν το έχω καταλάβει πάρα πολύ. Για τις τροπολογίες έχω να προσθέσω και μερικά πράγματα που χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλοί πολίτες ανησυχούν. Το ακούσαμε και στην ακρόαση και αυτά θα πρέπει να τα γράφει και η έκθεση, οι τροπολογίες. Ας πούμε, πολλοί πολίτες που ζουν σε άλλες χώρες από τις ε, πατρίδες τους έχουν ζητήματα. Μπορούν να υπογράφουν, δεν μπορούν να υπογράφουν στη συλλογή υπογραφών. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι οι πολίτες ε, μπορούν να υπογράψουν μια αναφορά ανεξαρτήτως αν είναι πολίτες της χώρας επίσης μετάφραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλε τι γλώσσε, αλλά υπάρχουν περιορισμοί προ του χαρακτήρε των μεταφράσεων. Αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο για τη μετάφραση. Και επίση θα πρέπει να ε, θυμόμαστε ότι όταν μεταφράζουμε από τη μία γλώσσα στην άλλη, μπορεί να είναι περισσότεροι χαρακτήρε, λιγότεροι. Κάθε γλώσσα δεν ε, ε, εκφράζεται με τον ίδιο ευσύνοπτο τρόπο. Μπορεί σε μία γλώσσα να χρειάζονται πολύ περισσότεροι χαρακτήρε για να πει το ίδιο πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και ε, τις μεταφράσεις για τα παραρτήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Και κάποιες ε, διευκρινήσεις ε, για τα πρακτικά και το κατά πόσο είναι νομικά παραδεκτό. Δεν ξέρουμε ξεκάθαρα τι εξαιρείται, τι είναι απαράδεκτο και για ποιο λόγο και προφανώς και ποιο είναι εκτός δηλαδή των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιες είναι πολιτικές ενέργειες που μπορεί να... Ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. The framework of the opinion provided Και ε, η νομική υπηρεσία του Κοινοβούλου μπορεί να μας διαφωτίσει. Τώρα για τη μερική καταχώρηση κάποιων πρωτοβουλειών θα πρέπει ε, πάλι να διευκρινιστεί το κείμενο και να μην υπάρχει καμία παρερμηνία αφησημία. Δηλαδή, ε, εάν ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλία είναι καλό, ανταποκρίνεται στα κριτήρια και είναι παραδεκτό, γίνεται μερικά αποδεκτή, μετά τι, τι συμβαίνει. Ένα τελευταίο, χωρί αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό. Αυτέ είναι οι βασικέ μου ανησυχίε και μελήματα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και στι νέε ε, διατάξει την προσβασιμότητα για την επιγραμμική συλλογή ε, υπογραφών. Να μην ε, εμποδίζεται κανένας λόγω κάποιων αδυναμιών ή ειδικών αναγκών. Αυτά έτσι πολύ σύντομα. Τα σχόλιά μου. Θα απαντήσει αμέσως ο η συγκεκριτή σας είπε, θα τα συμπεριλάβει στι τροπολογίε. Ωραία. Η Μπέτριθ Βεθέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα προφανώς να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Βαλένσα, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική εργασία. Και καλωσορίζω έτσι, με ευγνωμοσύνη την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πραγματικά βελτιώνει ουσιαστικά ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών κυρίως για να βελτιωθεί η δημοκρατία στην Ένωση γιατί αυτό είναι ο απότερος στόχος. Και οι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στη φάση καταχώρησης που τελικά ε, έχει γίνει κούρσα με τεμποδίων για να φτάσουμε σε κάτι που κανονικά έπρεπε να είναι πολύ απλό. Έχει τόσα προαπαιτούμενα, τόσο βαριά που δυσκολεύει. Εμείς οι φιλελεύθεροι ε, βλέπουμε ε, λοιπόν με ικανοποίηση κάποια στοιχεία ηλικία των 16 ετών, πολύ σημαντικό και για τους νέους να μπορούν να συμμετέχουν στη συμμετοχική δημοκρατία, τώρα που οι νέοι αρχίζουν να συμμετέχουν και σε άλλους κλάδους κοινωνίας και σε, στη ζωή την κοινωνική και στο άρθρο 4 για την ενημέρωση και τους διάβλους επικοινωνίας και παροχή συμβουλών. Πολύ συγκεκριμένη πρόοδος γιατί θα είναι βοήθεια αυτό για τους ε, πολίτες για να συλλέξουν τις απαραίτητες υπογραφές. Επίσης, ε, επιγραμμική πλατφόρμα, σημεία επαφή σε κάθε κράτος μέλος, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Και βεβαίως να διοργανώνεται διάσκεψη συνέχειας και παρακολούθησης για τις επιτυχείς ε, πρωτοβουλίες. Όλα αυτά θετικά και πρέπει να τα τονίσουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι το οποίο υπολοιπόμεθα. Η αρχική ιδέα στην πρώτη πρώτη έκθεση ποια ήταν. Και το είχαμε πει εμείς να χρησιμοποιούμε τα γραφεία που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Υπάρχει πρόταση να πηγαίνουν σε ορισμένα μέρη ε, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα έχουμε αρκετούς πόρους, αρκετούς υπαλλήλους, γραφεία. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πολλές φορές στην Επιτροπή Αναφορών. Εμείς είμαστε εδώ η μονοαπευθυντική θηρίδα στο Κοινοβούλιο για τους πολίτες. Το ίδιο θα πρέπει να είναι και ε, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Έχουμε επαγγελματίε εκεί, έχουμε ε, υπαλλήλου. Και ε, καλό θα ήταν να τους αξιοποιήσουμε πλήρως. Τώρα δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι πιο συγκεκριμένο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καλώς να ορίσει, αλλά θα πρέπει να αξιοποιούμε τους πόρους που υπάρχουν ήδη εκεί. Και είναι και εκπρόσωποι, ας πούμε, στις χώρες. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Αν θέλουμε πραγματικά να μεγιστοποιήσουμε την δημοκρατική δυναμική και το δυναμικό υπάρχουν κάποια στοιχεία από την νομοθεσία που δεν αποκρίνονται στις προσδοκίες ιδιαίτερα στην παρακολούθηση και στη συνέχεια που γίνεται στις παραδεκτές πρωτοβουλίες. Χρειάζονται οι πολίτες περισσότερη καθοδήγηση και προσανατολισμό. Όσοι έχουν υπογράψει οι διοργανωτές εδώ, το Κοινοβούλιο ε, μπορεί να έχει στρατηγικό ρόλο να διαδραματίσει και σε αυτή τη διάσκεψη θα πρέπει να πρωταγωνιστούμε πάντα στον πλευρό των πολιτών, έτσι ώστε η δουλειά που έχει γίνει να πιάνει τόπο και να δίνεται συνέχεια, έτσι, πιστή και δίκαιη. Θέλω να θυμίσω δύο πράγματα ακόμα. Εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε ή να μελετήσουμε το ενδεχόμενο αυτές οι πρωτοβουλίες που πέτυχαν, που πέρασαν όλα τα εμπόδια να, συζητούνται, να συζητούνται στην Ολομέλεια. Με ψήφισμα ή χωρίς. Πάντως εκεί να γίνει συζήτηση, εκεί που εδράζεται η εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει προτάσεις για τη σειρά με την οποία θα συζητηθούν και πότε. Αλλά δεν πειράζει να το συζητήσουμε, γι' αυτό δεν υπάρχει ολομέλεια. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα έρθουν στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, αλλά στην Ολομέλεια είμαστε όλοι παρόντες και εκεί μένει ο Ευρωπαίος πολίτης, εκεί κατοικεί στο ημικύκλιο. Τελευταίο. Για τη φάση της καταχώρησης επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντικατοπτρίζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του τελευταίου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πολύ πιο ρητή και να μας λέει για ποιο λόγο δεν δέχεται απορρίπτει δηλαδή ε, και να μας το ξεκαθαρίζει μια πρωτοβουλία. Έτσι θα βελτιώσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη με αυτό το αποτελεσματικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Ελιονόρα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την πρόταση που έχει κάνει σχετικά με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, ε, Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όσον αφορά τις ε, συνθήκες ε, πραγματικά έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέτει μια νομοθετική πράξη ε, και να περιμένει αυτό να στεφτεί από επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό με λυπεί πάρα πολύ. Αλλά βεβαίως και εμείς ή εγώ τουλάχιστον δεν είχα μεγάλο περιθώριο να καταθέσω τροπολογίες. Μπας περιπτώσει με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόταση που έκανε η δεύτερη συγγήτρια σήμερα η Ελίζα Λιρώνη, η οποία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με βάση το άρθρο 11 ε, έχουμε μια ε, νομική πράξη, legal act, η οποία νομοθετική με συγχωρείτε πράξη, αλλά μπορεί και να μην είναι νομοθετική. Είναι να προσπαθήσουμε να δούμε λιγάκι ε, ποια είναι τα περιθώρια που υπάρχουν, να προσπαθήσει το Κοινοβούλιο να ζητήσει μια μη νομοθετική πράξη, αλλά δεσμευτική εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό λοιπόν το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπας περιπτώσει... Ε... Εμείς ε, θα τοποθετηθούμε κυρίως σε τρία θέματα που ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο έχει σχέση με τις ε, διατάξεις σχετικά με την ΟΝΙΤΣΕ για να διασφαλίσουμε ότι η αξιολόγηση θα είναι διαφανής, αντικειμενική. Νομίζω ότι ακούσαμε πάρα πολλά κατά τη ακρόαση της ακρόασης, του διαμεσολαβητή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είναι δυνατό να υπάρξουν βελτιώσεις. Παραδείγματο χάρη έχουμε σκεφτεί ε, να υπάρχει ένα είδος ε, συμβούλου ελεγκτού με βάση αυτό που υπάρχει ήδη σήμερα όσον αφορά ε, το δικαίωμα ανταγωνισμού. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την αμεροληψία, τη διαφάνεια και μπορούμε ε, και να ε, επιδείξουμε και σεβασμό σε όλους τους άλλους ε, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να μπορούν να επιτύχουν μια τροποποίηση των συνθήκων με βάση αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο θα καταθέσουμε τροπολογίες. Και τέλος, ε, οι δημόσιες ακροάσεις οι οποίες κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να οργανώνονται από το Κοινοβούλιο, προφανώς με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και άλλων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων θα μπορούσε και αυτή να υπάρξει, γιατί κατά την άποψή μου ε, μερικές φορές απουσιάζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, δεν εκφράζεται η δική τους η άποψη, ακόμα και για επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών. Κατά την άποψή μου λοιπόν οι δημόσιες ακροάσεις ακόμα και μετά την παρουσίαση της ε, άποψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να κατατεθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονική περίοδο έτσι ώστε να είναι σαφές ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορούν να τοποθετηθούν οι πολίτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την ε, παρακολούθηση της υπόθεσης και αν δεν υπήρξε καμία συνέχεια να αναζητηθούν τα αίτια. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία προσέγγιση προς όφελος ε, του δημοσίου. Κατά τη δική μου άποψη δεν πρέπει να έχουμε εκπροσώπηση των ιδιωτών. Ε, αυτό που ενδιαφέρει κυρίω είναι ο σεβασμός του δημοσίου συμφέροντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Η κυρία Βαλένα. Ευχαριστώ. Και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κούνεβα που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. και έχει κάποια πράγματα για το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσει τον εισηγητή, τον κύριο Βαλέσα, για τις προτάσεις που έκανε και να υπενθυμίσει ότι ε, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα βήματα για τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας, τις πρωτοβουλίες ε, των πολιτών, οι οποίες ε, ε, τελικά αποτέλεσαν πονοκέφαλο κυρίως για τους διοργανωτές παρά οτιδήποτε άλλο. Και όπως είδαμε και εδώ στην Επιτροπή μας, αρκετές φορές υπήρχαν προβλήματα για τη συλλογή και την αναγνώριση των έγκυρων υπογραφών, το γεγονός ότι δεν διαφημίζονται οι πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει νομική αρρωγή και ορισμένες φορές από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δίνονται και απαντήσεις οι οποίες ήταν απαγοητευτικές. Ε, αρκεί κανείς να θυμηθεί την πρωτοβουλία για το νερό και όλα τα προβλήματα που είχε και το γεγονός ότι δεν απάντησε ε, τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οδήγησε και την ε, Ευρωπαία Διαμεσολαβητή να ξεκινήσει μια ε, διαδικασία για να δει ε, τι προβλήματα υπήρχαν. Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία λοιπόν να τροποποιήσουμε το παρελθόν και να γίνουν αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών ένα ισχυρό εργαλείο για την συμμετοχή των πολιτών και επίσης να μπορούμε να εγγυούμαστε την διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, υπάρχει νομική αρρωγή για τους διοργανωτές, ε, να μπορούν όλοι να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση και όχι μόνο στο διαδίκτυο ε, και να εξηγούν και τους λόγους για τους οποίους ε, απορρίπτεται δράση σε μια πρωτοβουλία παρά το γεγονός ότι ορισμένες φορές είναι δεόντως αιτιολογημένη και τελικά απορρίπτεται. Απαιτούμε μεγαλύτερη διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών και αυτό φυσικά νομίζω ότι συνοψίζει όσα ελπίζουμε να έχουμε με αυτή τη γνωμοδότηση και τη γενική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπόργαρτ, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσουμε ε, που είσαστε σχεδόν όλη μέρα εδώ. Ελπίζω να μην ήταν πάρα πολύ δύσκολο για σας, είστε πολύ εχθρικό το κλίμα και να μας ξανάρθετε χαμογελαστό. Βεβαίω θα ξανάρθω. Εκτός του ότι είναι η δουλειά μου και πληρώνομαι γι' αυτό. <laughs> Μ' αρέσει κιόλα. Όχι καθόλου εχθρικό δεν ήταν. Τα περισσότερα από τα σημεία αυτά τα έχουμε αντιμετωπίσει με τον αλφαβήτα τρόπο. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι για τη μετάφραση των πρωτοβουλειών. Έχουν αυξηθεί οι χαρακτήρες ε, ε, από 800 σε 1100. Υπάρχει λόγος που περιορίζουμε τους χαρακτήρες τους υπογραφικού. Ε, γιατί θα πρέπει να χωρέσει μία σελίδα το κείμενο. Εξού και οι υπογραφές περιορίζονται σε τρεις. Υπάρχει και το θέμα των παραρτημάτων, προστασία δεδομένων κλπ. Θέλουμε να έχουμε μία σελίδα που να μπορεί κάποιος να τη διαβάζει ε, και στο ίντερνετ και στο χαρτί. Θα σας δώσουμε περισσότερες ε, λεπτομέρειες αν θέλετε για τα τεχνικά ε, ζητήματα για να κατανοήσουν όλοι τι προτείνουμε. Αν θέλετε να είμαστε πιο γενναιόδοροι υπάρχει δυνατότητα αλλά δεν χωράει σε μια σελίδα και δεν θα είναι τόσο φιλικό προς το χρήστη αυτό το σχήμα. Εξού και οι τρεις υπογραφές. Και όσο πιο μικρή είναι η γραμματοσυρά, τόσο πιο δύσκολο είναι για το χαρτί, που δεν είναι επιγραμμικά ε, πάντα τα υποστρώματα. Υπάρχουν και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας κλπ. Ξέρω ότι ορισμένοι θέλουν να πούμε τι εξαιρείται ρητά να το γνωρίζουν από τις δικές μας αρμοδιότητες και εξουσίες. Είναι μεγάλη διακριτική ευχέρεια, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να το κάνει και μετά ε, μας κατηγορείται. Αλλά αν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής, υπάρχει ήδη. Είναι πολλαπλές οι ε, πρωτοβουλίες παντός είδους και εάν ο ορισμός και το πεδίο εφαρμογή έχει οριστεί με πάρα πολύ στενή έννοια, τότε το δικαστήριο κατά την προσφυγή θα είναι υποχρεωμένο να πει ότι είναι εκτός πεδίου. Το άρθρο 288 είναι, αν δεν απατώμε από τη συνθήκη, έτσι, εδώ, ε, έχω ξεκάθαρο δηλαδή μπορούμε καλόπιστα ε, ε, να περιορίζουμε ακόμα περισσότερο το πεδίο και Κινδυνεύουμε να το κάνουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ γενναιόδορη ε, στην πράξη στις αποφάσεις της. Στο μέλλον, αν πάρουμε μια απόφαση να αποκλείσουμε κάτι, πάλι θα υπάρχουν γκρίνιες και καταγγελίες και θα μας κατηγορούν ότι στο παρελθόν ήμασταν πιο γενναιόδοροι. Και θα έρχεται το δικαστήριο να μας θυμίσει τη δική του νομολογία. Καλές είναι οι βελτιώσεις, αλλά στη νομική αποτίμηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, προσεκτική ε, η προσπάθεια αυτή και επί της ουσίας νομικής δηλαδή, γιατί κινδυνεύουμε να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής υπερβολικά. Και αυτό μας απασχολεί βεβαίως. Συνέχεια στο Κοινοβούλιο έχω σημειώσει εδώ, προφανώς είμαστε στα χέρια σας, αλλά ως πολίτης φυσικά με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Οτιδήποτε μπορεί να, αφήσει, να ε, διατηρήσει την ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό ε, θα ατύχει ευνοϊκής υποδοχής από τους πολίτες. Αλλά να μην το παρακάνουμε γιατί σε τελική ανάλυση είναι διοικητική η αρμοδιότητα δικιά μας, όχι πολιτική. Α, υπήρξε και ένα άλλο θέμα. Α, θα γίνει. Ακρόαση όχι. Εγώ έχω διατελέσει ε, σε γραφείο επιτρόπου ε, ε, θέματα ανταγωνισμού, αλλά είναι περιορισμένος ο ρόλος μας. Είναι διαμεσολαβητικός, δεν έχουμε... Πώς να το πω, να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο με μια άλλη αρχή ε, αυτό που προσπαθούμε να απλουστεύσουμε. Δεν εξυπηρετεί το στόχο ούτε ως προς την ταχύτητα και τη ροή της διαδικασίας. Και μετά πάλι θα κληθεί να λογοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το μόνο που θα κάνουμε θα, έχουμε και έναν επιπλέον υπάλληλο αρμόδιο για την ακρόαση. Είχαμε που είχαμε ένα δίμηνο, αλλά τελικά θα, θα αποδειχθεί πολύ λίγο αυτό. Δεν είναι όλα προφανή και αυτονόητα. Πολλές φορές ε, οι νομικοί ε, δεν συμφωνούν. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα δωμάτιο τρεις νομικούς να συζητήσουν για ένα πρόβλημα, θα, με τρεις απόψεις, βγαίνοντας από το δωμάτιο θα έχουν τέσσερις απόψεις. Έλεγχος γίνεται, σε μία από το σώμα των επιτρόπων. Εμείς περιοριζόμαστε στο νομικό έλεγχο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με την καταχώρηση. Και υπάρχει λόγος που έχει επιλεγεί συγκεκριμένη διατύπωση και στη νέα ε, πρόταση. Όσο το φουσκώνουμε αυτό το θέμα όμως, τόσο θα ε, επιβαρύνει τη διαδικασία. Το τελευταίο διάστημα απορρίφθηκε μία ε, πρωτοβουλία, ε, το τίτλο Stop Brexit. Με Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Γιάρεκ, θες να προσθέσεις τίποτα, κύριος Παλένσα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο ε, σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία για τη δική μας την Επιτροπή. Υπάρχει αυτό το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να περάσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι πολύ σημαντικό ε, να τα κάνουμε όλα σωστά. Ε, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτά που μας είπατε σήμερα ε, όταν θα έχουμε τις τροπολογίες. Τότε θα, τα, τοποθετηθώ εκτενώς, αλλά ήδη τώρα θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της φυσικής επαφής. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά σήμερα παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε κινητό, ούτε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Είναι δύσκολο λοιπόν για αυτούς να έρθουν σε επαφή με γραφεία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα ε, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, να προσφερθούν για αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ ε, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Αυτό μπορεί να γίνει προαιρετικά, να προσφέρουμε πακέτα ενημέρωσης για όσους ενδιαφέρονται για ε, τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα ε, και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει και δυνατότητα να υπάρχουν σημεία επαφής. Ξέρω ότι συμφωνούμε για τα περισσότερα θέματα και όταν θα δούμε συγκεκριμένα τις τροπολογίες είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε μία μορφή σε αυτή τη γνωμοδότηση με την οποία θα συμφωνούμε όλοι το δικό σας το γραφείο, γιατί να μην το κάνουμε σημείο επαφή. Ήδη είναι, λέει ο κύριος ε, ε, ε Σήμερα λοιπόν είχαμε την εξέταση αυτής της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης ε, στις 3 ε, η ώρα, 3 Μαρτίου, είναι καταληκτήρια ημερομηνία, 24 Απριλίου θα ψηφίσουμε και στις 24 Μαΐου την Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Θα τα πούμε αύριο. Στις 9 η ώρα οι συντονιστές και οι υπόλοιποι στις 10.30.